Καλημέρα σα, Πάρτε, ελάτε στι θέσεις σα. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής. Νομίζω ότι ο κύριος Σουμπιόλσκι ήταν κάποιο από όσου έλαβαν την πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτή τη ακρόαση σήμερα το πρωί. Θα έρθει μαζί μα. Λοιπόν, αντικείμενο... Ε, το αντικείμενο είναι η ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ε, δημοκρατίας στην, ε, στους κόλπους της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Και κάνουμε αυτή τη συναντρία σε μια δύσκολη στιγμή της ε, διαδικασίας αυτής που συνδέεται, δυσκολία που συνδέεται με τον πόλεμο της Γάζας και τελμάτωσης. Και δεν παρίσταται ο εκπρόσωπος ε, της Αιγύπτου στο... σήμερα το πρωί ξέρετε ότι έχουν, οι συνεδράσεις στο πλαίσιο αυτό έχουν παγώσει. Θα εμβαθύνουμε αυτό στη συζήτηση αυτή δίνοντα το λόγο στην κυρία Ναπολιτάνο η οποία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει αναλάβει μια έκθεση της οποίας η ψηφοφορία έχει αναβληθεί ακριβώς λόγω της κατάστασης στη Γάζα αλλά έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου εάν δεν απατώμε και στο ψήφισμα το οποίο ε, προτείνει ε, επιμένει πάρα πολύ στην ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, ευρω, ευρωπεριφερειακή μεσογειακή κλίμακα και αναφέρεται στο μηχανισμό ο οποίος προέρχεται από τη δικασία της Βαρκελόνης για τον οποίο έχουν συσταθεί ορισμένα εργαλεία, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά, εργαλεία για την ενίσχυση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας και οι νέες διατάξεις που συνδέονται με την Ευρωμεσογειακή Ένωση και που εστιάζουν κυρίως στα μεγάλα προγράμματα σε περιφερειακή κλίμακα. Και θα δούμε και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιες είναι οι καινοτομίε, ούτω ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ούτω ώστε να πετύχουμε το στόχο αυτό που μας συνενώνει εδώ σήμερα. Λοιπόν, για την ε, παρουσίαση του θέματος αυτού, συγγνώμη, θα δώσουμε το λόγο στην Πασκαλίνα Ναπολιτάνο και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον ε, Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης ΡΕΛΕΞ, τον κύριο Μεσόν, ο οποίος βρίσκεται εδώ από το Κέντρο για τις ε, Μελέτες της Ευρωμεσογειακής Πολιτικής και ένα μέλος εκτελεστικής επιτροπής του Ευρωμεσογειακού Δικτύου και της ε, μη κυβερνητική ε, πλατφόρμας Euromed. Κυρία Πασκολίνα Ναπολιτάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως υπενθυμίσατε κι εσείς, την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες θα ψηφίσουμε την έκθεση του Κοινοβουλίου με θέμα την Ένωση για τη Μεσόγειο. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κάποιο αδιέξοδος εξελίξης στην ανάπτυξη των νέων φορέων που προβλέπονται από τη Συμφωνία. Και νομίζω ότι ως συνήθως το Κοινοβούλιο θα δώσει μια συνεισφορά επικοδομητική με σκοπό να αναπτύξουμε μια συνεπή πολιτική, μια συνεκτική πολιτική. Εμείς οι ίδιοι έχουμε ήδη υπογραμμίσει κάποια στοιχεία της περιπλοκότητας ε, σε ό,τι αφορά τη σχέση Ευρωπαϊκής τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και των επιμέρου ακόμα κρατών μελών με τι υπόλοιπε μεσογειακές χώρες. Μπορώ να πω ότι ο χώρο αυτό έχει μια μεταβλητή γεωμετρία. Έχουμε διάφορα εργαλεία τα οποία συνυπάρχουν. Και συχνά δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να τα ενσωματώσουμε σε ένα συνεκτικό πλαίσιο όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω ακριβώς ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο θα περιλαμβάνει και θα αντικαθιστά τελικά τη διαδικασία της Βαρκελόνης και θα περιλαμβάνει τις νέες ε, πρωτοβουλίες που προέβλεψε η Σύνοδος Κορυφής ε, του Παρισιού στις 14 Ιουλίου και όσα αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών στη Μασαλία. Δηλαδή, ενώ πριν χρησιμοποιούσαμε την έκφραση διαδικασία της Βαρκελόνης, Παύλα, Ένωση για τη Μεσόγειο, τώρα αυτή η έκφραση, Ένωση για τη Μεσόγειο, αντικαθιστά την προηγούμενη έκφραση. Όλα αυτά δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα, γιατί το κεκτημένο της Βαρκελόνης παραμένει. Ξέρουμε ότι αυτό το πλαίσιο, αυτή η συμφωνία πλαίσιο που ενώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες ε, μεσογειακές χώρες βασίζεται σε ένα έγγραφο που προβλέπει τους διαβόητους τρεις πυλώνες, αλλά προβλέπει επίσης και ένα σύστημα χρηματοδότησης των πρωτοβουλειών και των προγραμμάτων που βασίζονται 100% στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μιλάμε τώρα για περιφερειακά προγράμματα, υπερπεριφερειακά προγράμματα και διμερή προγράμματα. Μην ξεχνάμε επίσης και την πολιτική γειτονίας που, που παραμένει ε, με τις χώρες ε, του Νότου, που θεωρείται όμως διμερής πολιτικής, που βασίζεται σε σχέδια δράσης Υπάρχουν κάποια στοιχεία ρεσιμότητας σε ό,τι αφορά δηλαδή το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημιουργία ενός κράτους δικαίου. Αυτή η πολιτική λοιπόν δεν εξαλείφεται, παραμένει. Τώρα, τι προσθέτει τότε η Ένωση για τη Μεσόγειο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο προσθέτει καταρχάς την αρχή ότι πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένες οι πολιτικές. Οι πολιτικές πάβουν να είναι αφηρημένες. Δηλαδή, μέσα από την, μέσω της ιδέας των νέων προγραμμάτων και της ιδέας της ε, γραμματείας που τα διαχειρίζεται, που τα δρομολογεί και τα διαχειρίζεται, δίνεται έμφαση σε μια εδαφική πολιτική μιας μεγαλύτερης ε, δαφικής ολοκλήρωσης, εδαφική συνοχής σε πολυμερές επίπεδο που λαμβάνει η χώρα στη Μεσογειακή Λεκάνη, στο Μεσογειακό χώρο. Τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε δηλαδή για οικονομική ολοκλήρωση, περιβαλλοντική ολοκλήρωση, διαφορετική ολοκλήρωση. Με σχέδια δράσης και συγκεκριμένα προγράμματα στο Μεσογειακό χώρο. Η χρηματοδότηση για αυτές τις πρωτοβουλίες δεν είναι αποκλειστικά δεν είναι αποκλειστικά ευρωπαϊκή, αλλά είναι διμερής. Και εμπεριέχουν την ιδέα της συμμετοχής των χωρών εταίρων του Νότου. καθώς και τα, τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών, τον κοινοτικό προϋπολογισμό βέβαια προφανώς, καθώς και ιδιωτικά κονδύλια, τα οποία είναι ευπρόσδεκτα. Φυσικά, όταν κάποιος ε, ρωτάει γιατί δεν μπορεί η Κομισιόν να διαχειριστεί όλη αυτή η διαδικασία η απάντηση βρίσκεται και στη φύση της χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται τον ε, κοινοτικό προπολογισμό και όχι ιδιωτικά κονδύλια ή κονδύλια άλλης φύσεως. Η Ένωση για τη Μεσόγειο δημιουργεί για κάποιους θεσμούς για τον πολιτικό διάλογο, που μέχρι στιγμής η διαδικασία της Βαρκελόνης δεν είχε προβλέψει, δεν είχε κωδικοποιήσει όπως παραδείγματος χάρη την έννοια της συμπροεδρίας. Που αυτή τη στιγμή την, την έχει αναλάβει η Αίγυπτος από τη μία φορά. Από την πλευρά της Ευρώπης τα πράγματα είναι πιο συγκεχημένα, γιατί από ό,τι φαίνεται η Γαλλία του Σαρκοζή συνεχίζει τη συμπροεδρία αλλά η συνθήκη προβλέπει άλλα πράγματα. Επομένως, το Κοινοβούλιο θα παρουσιάσει μια τροπολογία στο Συμβούλιο για να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνέχεια σε αυτή την εκπροσώπηση της Ευρώπης μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και να δώσει στην Ένωση για τη Μεσόγειο μια μεγαλύτερη σταθερότητα και μια σαφέστερη ταυτότητα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Υπάρχει όμως και η συγκέντρωση των Υπουργών Εξωτερικών όλων των χωρών της ανάσχετης Μεσόγειο και των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και βεβαίως και η γραμματεία που θα έχει πιο λειτουργικό ρόλο. Αυτό είναι θετικό. Βέβαια το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει και τις αντιφάσεις πέρα από τα θετικά στοιχεία. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη διαδικασία η οποία δημιούργησε μια πραγματική εταιρική σχέση. Δηλαδή, οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες του Νότου συνεργάζονται και δημιουργούν κάποιους θεσμούς. Αυτό είναι θετικό. Θυμάμαι στην προηγούμενη θητεία σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική γειτονία, εμείς είχαμε το επιμείνει προς το Συμβούλιο και προς το, την Κομισιόν να δημιουργηθούν θεσμοί, φορείς. Γιατί δεν γίνεται να ασκήσουμε πολιτική χωρίς θεσμούς. Η Σύνοδος Κορυφής του Παρισιού μιλάει για θέματα κάτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά είναι σαφές ότι αυτοί οι θεσμοί, η Συμπροεδρία, η Σύνοδος Κορυφής των αρχιών Κρατών και Κυβερνήσεων και οι συνεδριάσεις Υπουργών Εξωτερικών δεν θα συζητάνε κατά κανόνα τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ακριβώς γι' αυτό η Amnesty International, το Ινστιτούτο του Καΐρου, η Human Rights Watch και η Euromed Rights έστειλαν μία επιστολή που υπογραμμίζουν αυτό το στοιχείο. Επομένως, ο πολιτικός διάλογος δεν επικεντρώνεται από ό,τι φαίνεται σε αυτά τα θέματα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ως Κοινοβούλιο επικρίναμε το κριτήριο αυτό που οδηγεί το Συμβούλιο και εν μέρη την Κομισιόν στο να προτείνει την αναβάθμιση στις σχέσεις με κάποιες χώρες, ιδίως με το Ισραήλ και το Μαρόκο, όπου αυτά τα θέματα του κράτους δικαίου και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας ξεχνιούνται. Είναι αλήθεια βέβαια, το 2008 το Ισραήλ αύξησε κατά 60% την προσπάθεια απικιοποίησης της δυτικής όχθης. είναι ένας κόλαφος για το διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό το ξεχνάμε στην αξιολόγηση. Επίσης, το Μαρόκο, που είναι μια ενδιαφέρουσα χώρα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά υπάρχει μια κρυφή σύγκρουση εκεί, της Δυτικής Σαχάρας. Η λύση σίγουρα είναι περίπλοκη και τίθενται προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μην ξεχνάμε την περασμένη εβδομάδα μία αντιπροσωπεία μας πήγε επί τόπου και είδε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Ιδίως ό,τι αφορά τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά τη ζωή αυτής της μειονότητας που είναι απίστευτα δύσκολη. Όλα αυτά ξεχνιούνται εντελώ. Δεν αναφέρονται όταν γίνεται λόγος για upgrading, για αναβάθμιση των σχέσεων. Συμμετείχα μαζί με άλλους συναδέλφους σε μια συνάντηση με κάποιους υπαλλήλους της Κομισιόν που διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή την Συμφωνία Σύνδεσης με τη Λιβύη. Αυτοί οι υπάλληλοι της Κομισιόν μας είπαν ότι το πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ξεκινάει με την ε, περίφημη φράση «Συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες και το, την ιδέα του κράτους δικαίου». Εμείς αρχίσαμε γελάμε. Ε, μην το πείτε καλύτερα. Ε, πείτε κάτι πιο τίμιο. Ότι μας ενδιαφέρει να έχουμε μια σχέση με τη Λιβύη ανεξάρτητα από το κράτος δικαίου και την εξέλιξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου. Γιατί είναι γελία να λέμε αυτά τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα εργαλεία, χάνεται κάθε έννοια, ας πούμε, γύρω από αυτά τα θέματα. Καλύτερα να πούμε πιο τίμια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να αλλάξει. Δεν προτίθεται να θέσει ως προϋπόθεση για την, τις αναπτυξιακές σχέσεις τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ή αν θέλουμε να το κάνουμε, ας είμαστε πιο αξιόπιστοι. Θα πρέπει να έχουμε εργαλεία πιο αξιόπιστα. Μέχρι στιγμής είδαμε ότι η ρήτρα αυτή που έχουμε στο δεύτερο σημείο των συμφωνιών σύνδεσης ποτέ δεν παρήγε μια καταγγελία από πλευρά Ευρώπη και η ίδια η προϋπόθεση που προβλέπεται στα σχέδια δράσης, κάτι αντίστοιχο, δεν οδήγησε σε καμία ουσιαστική αλλαγή σε καμία εξέλιξη. Και αυτό προκύπτει και από πρόσφατες μελέτες. Από, πολλούς, από πολλούς διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Αλλά προκύπτει και από τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Επομένως, καλό είναι να γίνει ένας απολογισμός τίμιο είναι να γίνει σε απολογισμός. Για να δούμε τι εργαλεία θα πρέπει να έχουμε στο μέλλον. Οι προϋπόθεσεις αυτές που βάζουμε μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις καταστάσεις. Έχουμε αμφιβολίες. Η ρήτρα του δεύτερου εδαφείου των συμφωνιών δεν οδήγησε σε τίποτα. Άρα έχει νόημα αυτή η ρήτρα. Όλοι γνωρίζουμε το εξή ότι η ευρωπαϊκή εμπειρία μας λέει ότι μόνο η πλήρης ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μας οδήγησε σε ουσιαστικές αλλαγές στις χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις. Αν δεν υπάρξει πλήρης ολοκλήρωση, δηλαδή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εμπειρία τι μας λέει, ότι οι χώρε αυτές θα εξελιχθούν προ τη δική του κατεύθυνση, όπως τη Λατινική Αμερική, που έγιναν τόσες αλλαγέ που δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Αλλιώ η Ευρώπη και τα όργανά της, τα εργαλεία τη κτλ. καθορίζουν ελαχιστότατα αυτές τι εξελίξεις. Εν τούτης, εμείς έχουμε μία ευρωμεσογειακή κοινοβουλευτική συνέλευση. Δημιουργήσαμε αυτή τη συνέλευση δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας της Βαρκελόνης. Ίσως θα πρέπει να δούμε πώς θα ενταχθεί τώρα αυτή σε αυτό το νέο σχήμα Ένωση για τη Μεσόγειο. Υπήρχαν, υπήρξαν και άλλες εμπειρίες με την Ανατολική Ευρώπη, όπου είχαμε Έχουμε δυσκολίες αυτές τις αλλαγές να τις εφαρμόσουμε στον αραβικό κόσμο. Γιατί πιστεύουμε ότι οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες δεν έχουν τάσεις ε, δημοκρατικές αντίστοιχες με τις δικές μας ευρωπαϊκές τάσεις. Και επομένως δεν διανόμαστε καν ότι υπάρχει μια περίπτωση εξέλιξης ε, της κατάστασης, περίπτωση εξέλιξης της σχέσης μας. Τι εννοώ, ότι αυτές οι χώρες, καλώς ή κακώς, με κάποιες εξαιρέσεις, συμμετέχουν στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας σε κάποιες χάρτες όπως του ΟΗΕ, σε κάποιες διεθνείς συμβάσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από εκεί, από αυτή τη συμμετοχή τους, για να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές κοινέ αξίες μας και όχι αυτά τα αφηρημένα που καθόμαστε και λέμε, όπως κάνουμε με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θεωρούμε ότι η βάση είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, αν το σκεφτούμε καλά το θέμα, με αυτές τις χώρες δεν έχουμε καμία κοινή νομική πράξη που μας πείθει ότι έχουμε κοινέ αξίες. Γιατί η ρήτρα του εδαφίου 2 των συμφωνιών είναι μάλλον ευρωπαϊκής έμπνευσης. Δηλαδή οι χώρε αυτέ δεν θέλουν δική τους αυτή η ρήτρα. Διαισθάνονται ότι όταν το Κοινοβούλιο εκφράζεται μέσω κάποιων ψηφισμάτων προτάσεται αυτή η ρήτρα, αλλά τελικά το Κοινοβούλιο διαψεύδεται από τη στάση του Συμβουλίου που τους λέει «Ε, αφήστε τώρα το Κοινοβούλιο, μερικές φορές έχουν ανάγκη έτσι να τα βγάζουν από πάνω τους αυτά αυτό το βάρος». Εμείς θέλουμε να επιλύσουμε μαζί σας άλλα προβλήματα. Με εμά έχετε να κάνετε. Ίσως θα έπρεπε να βασιστούμε σε κάτι το οποίο πραγματικά συμμεριζόμαστε εμείς και οι χώρες αυτές. Για να δημιουργήσουμε έτσι μια αίσθηση ευθύνης ε, και από αυτές τις χώρες εταίρους ε, για αυτές τις σχέσεις. Σε αυτή την έκθεση θέλουμε λοιπόν να υπάρξουν εργαλεία πιο στενάρα, ε, πιο ουσιαστικά, πιο απτά, ε, μέσω των οποίων θα εκπροσωπείται η κοινωνία των πολιτών. Να υπάρχουν και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Ζητάμε να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις συνεδριάσεις του Μεσογειακού Δικτύου της Κοινωνίας των Πολιτών. που εκφράζει εδώ και πολλά χρόνια την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα αυτή πρέπει να τη δούμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα, να τη λάβουμε υπόψη μας με μεγαλύτερη σοβαρότητα. Σε πολλές από αυτές τις χώρες υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν οργανώσεις των επιχειρηματιών, υπάρχουν οργανώσεις των γυναικών. Θα πρέπει να βοηθήσουμε για να αποκτήσουν μια δομή πιο συγκεκριμένη. Ζητάμε, παραδείγματο χάρη, να δημιουργηθεί μια οικονομική Επιτροπή. Μεσογειακή. Παραδείγματο χάρη, είδαμε ας πούμε ότι ο επιχειρηματικός τους κόσμος κινείται, είναι πολύ πιο μπροστά από ότι η πολιτική τους στις περιφερειακές σχέσεις. Ενώ η πολιτική είναι πολύ πιο εθνικιστές, αν θέλετε, σε αυτές τις χώρες. Οι οργανώσεις των γυναικών σε πολλές από αυτές τις χώρες ε, έχουν βοηθήσει ε, να αλλάξει και η νομοθεσία. Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να δώσουμε φωνή και βήμα σε αυτές τις οργανώσεις που υπάρχουν στις κοινωνίες αυτών των χωρών. Η κατάσταση πραγματικά είναι αντιφατική σε αυτές τις χώρες. Αυτή τη στιγμή όλοι οι θεσμοί της Μεσογειακής, της Ένωσης για τη Μεσόγειο βρίσκονται σε φάση έτσι, παγώματος λόγω της Γάζας. Το Κοινοβούλιο θέλει να βοηθήσει για να ξαναρχίσουμε την πορεία. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να κινηθούν και, τα, και οι θεσμοί της α, κοινοβουλευτικής συνέλευσης, που μέχρι στιγμής έχουν δώσει σημαντικά ωφέλη. Ευχαριστούμε πολύ Πασκουαλίνα που δεν ε, χειρίζεται, δεν διαθέτει μια ξύλινη γλώσσα όπω άλλοι και έχει πολλέ ιδέε ούτω ώστε να δώσει μια όθηση σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα έχει το λόγο η Κομισιόν, ο κ. Φλάντε Μοράλ, για να μα ε, παρουσιάσει την κατάσταση και τους μηχανισμούς που μπορεί να κινητοποιήσει η Κομισιόν για να είναι πιο αποτελεσματική στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την υποεπιτροπή σας και την πρόεδρο, την κυρία Φλόδρο, για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Ναπολιτάνο για την προετοιμασία της τελικής έκθεσης για την διαδικασία της Βαρκελόνης για την ευρωμεσογειακή διαδικασία που θα συζητηθεί όπως ακούσαμε στις 18 Φεβρουαρίου αλλά και για τα όσα μόλις είπε. Ανέφερε κάποια ζητήματα που μας απασχολούν. Τον Ιούλιο του 2008 στο Παρίσι είχαμε 43 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μεσόγειο που συμφώνησαν να βασιστούν στα επιτυχή στοιχεία της διαδικασίας Βαρκελόνης μέσω πρώτων της αναβάθμισης των σχέσεών τους, δηλαδή να είναι στο επίπεδο σύνοδων κορυφής. Δεύτερον, μέσω της σύστασης θεσμικών οργάνων και τρίτον μέσω της παροχής συγκεκριμένων απτών πλέον εκτιμάτων για τους πολίτες, κάτι το οποίο έλειπε στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσόρισε τα αποτελέσματα της Συνόδου και συμμετείχε ενεργά στην ε, διακήρυξη, στη σύνταξη της διακήρυξης, στην οποία κατέληξε η Σύνοδος. Νομίζουμε πως είναι ένα σημαντικός τρόπος πρόοδου της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Η τελική διακήρυξη μιλάει για μια κοινή δέσμευση για τη δημοκρατία και τον πολιτικό πλουραλισμό μέσω της διεύρυνσης συμμετοχής στην πολιτική ζωή και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημείωσα αυτά τα οποία είπε η κυρία Ναπολιτάνου για τις κοινέ αξίες, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να σημειώσουμε είναι πως αυτός ο πολιτικός στόχος είναι ίδιος με αυτόν της διαδικασία της Βαρκελόνης. εμείς στην Επιτροπή αναζητούμε τρόπους να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε διάφορα επίπεδα. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας και της ε, Ένωσης για την Μεσόγειο και πρέπει να σημειώσουμε πως αυτή η Ένωση βασίζεται στην προϋπάρχουσα ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση, αρχές τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Όπως σας διάβασα μόλις, το πολυμερές αυτό πλαίσιο έχει στόχους όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά δεν έχει μηχανισμούς, αν και κάποιες δράσεις αναπτύσσονται. Η εμπειρία μας δείχνει πως ε, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι το διμερές πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας με βάση τις συμφωνίες σύνδεσης. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα που ανέφερε και η κυρία Ναπολιτάνο, η περίπτωση του Μαρόκου. Μια χώρα που ήδη βρίσκεται στην επόμενη φάση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Να σας πω πρώτα απ' όλα πως η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας δεν είναι εντελώς διμερής υπόθεση, εφόσον οι στόχοι είναι κοινοί, μιλάμε για μία σύγκληση προς κάποιες αξίες, ε, προς κάποιες οικονομικούς στόχους και προς το επίπεδο διαβίωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παρόμοια είναι και τα μέσα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα στην περίπτωση του Μαρόκου, που είναι ίσως η πιο προχωρημένη περίπτωση νέων στόχων, της νέας αυτής φάσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Εάν δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα βλέπουμε πως έχουμε προχωρήσει παραπέρα καθώς θέλει να συγκλίνει το Μαρόκο. Έχουμε τη φιλοδοξία του να υπογράψει κάποιες συμβάσεις Συμβουλίου της Ευρώπης. Οπότε έχουμε κάποια βήματα προς την κατεύθυνση που θέλουμε. Τα σχέδια δράσης ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας αφορούν δεσμεύσει στον πολιτικό διάλογο, τη μεταρρύθμιση ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες όπως ε, η ελευθερία της έκφρασης, ε, του συνεταιρίζεστε, τα δικαιώματα των γυναικών και η δικαιοσύνη. Έχουμε δηλαδή συγκεκριμένους στόχους με βάση την κάθε συμφωνία. Έχουμε ενισχύσει τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις μεσογειακές ε, χώρες στις ε, υποεπιτροπές με την ε, Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο, την Ισία, Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ. Και στοχεύουμε να επεκτείνουμε το έργο αυτών των υποεπιτροπών. Προτείναμε ήδη την πρώτη μας συνάντηση με την Παλαιστινιακή Αρχή και το ίδιο θα γίνει με το Ισραήλ. Οι συνεδριάσεις αυτές ε, εξετάζουν την πρόοδο ή τιμή πρόοδο αναλόγως όσον αφορά την εφαρμογή των δεσμεύσεων των σχεδίων δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Τον Απρίλιο που μας πέρασε έκανα μια γενική αξιολόγηση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, γειτονίας. Είδαμε κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Μια άλλη ποιοτική αλλαγή στις μεθόδους εργασίας μας είναι πως ε, συμβουλευόμαστε τις ΜΚΟ στις ε, αρμόδιες αυτές υποεπιτροπές. Επίσης, υποστηρίζουμε με τον κοινοτικό προϋπολογισμό την τοπική κοινωνία των πολιτών, κυρίως μέσω του ευρωπαϊκού μέσου που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και μέσω, μέσων της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Και βεβαίως στοχεύουμε και στην παροχή υπηρεσιών για όλα τα οικονομικά, κοινωνικά και λοιπά δικαιώματα. Σημειώνουμε την πρόοδο πύχη στη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, ε, την διακυβέρνηση του τομέα, πράγματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά η εικόνα είναι μεικτή όσον αφορά το σεβασμό των ε, ατομικών ελευθεριών, τα πολιτικά δικαιώματα κτλ. Σε κάποιες χώρες έχουμε σοβαρούς λόγους ανησυχίας Υπάρχουν προβλήματα με τη θανατική ποινή, δεν υπάρχει η ελευθερία του συνεταιρίζεστε, περιορισμοί στη χρηματοδότηση μη καπαόμικρων, περιορισμοί της δράσης ε, υπηρεσιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλείσιμο μη καπαόμικρων, περιπτώσεις ε, δυσφημίσεως, ε, βασανιστήριων, παραβίαση των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών. Επίσης το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις εκλογές στις περισσότερες χώρες δεν ε, συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ανθρώπινα δικαιώματα και στην κατάσταση της δημοκρατίας στις μεσογειακές χώρες. Πέραν από τις συγκεκριμένες υποεπιτροπές, εμείς θίγουμε αυτά τα ζητήματα σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού διαλόγου με τις χώρες αυτές. Επιπλέον, εκφράζουμε τις ανησυχίες μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αμελιώδεις ελευθερίες μέσω των διπλωματικών διάβλων, υπενθυμίζουμε στους εταίρους μας τις διεθνείς τους δεσμεύσεις σύμφωνα και με τα σχέδια δράσης της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Επίσης η πολιτική μας φαίνεται και με τον τρόπο σύνταξης των ε, εγγράφων στρατηγικής αναχώρα για το 2007-2013 δίνεται βάρος στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αμελιώδεις ελευθερίες. Παραδείγματος χάρη, δική προτεραιότητα στα ενδεικτικά προγράμματα 2007-2013 προέβλεπε υποστήριξη στην εξέλιξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την προτεραιότητα και μετά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Μα έρθω τώρα στην πολυμερή αυτή προοπτική που είναι ο στόχος μας σήμερα. Το πολυμερές πλαίσιο εμείς θεωρούμε πως ε, μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτές τις περιφερειακές προκλήσεις όπως π.χ. η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών. Η Κομισιόν βρίσκεται σε έναν διάλογο με μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε πολλούς τομείς. Θεωρούν πως η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ενισχυθεί και οι δυνατότητές της μέσω της αλληλεπίδρασης με κυβερνήσεις και κοινοβούλια. Γι' αυτό, παραδείγματο χάρη, η Κομισιόν υποστηρίζει την πλατφόρμα ΜΚΟ, την Ευρωμεσογειακή, και άλλα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών μέσω του τοπικού φακέλου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Ο στόχος μας εδώ πέρα λοιπόν είναι να συνεχιστούν αυτές οι εξελίξεις μέσω ε, του προγράμματος ε, ανάπτυξης ε, αστικής και διαλόγου για να υπάρξουν μακροπρόθεσμα τέτοια σχεδιαστική ανάπτυξης. Επίσης, μπορούμε να δούμε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως παραδείγματο χάρη ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η εμβάθυνση του περιφερειακού διαλόγου, με το να μοιραζόμαστε βέλτιστε πρακτικές στον τομέα των εκλογών, όχι μόνο με του εταίρου μα. Το συζητάμε και με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Η μεταρρύθμιση στον τομέα του πολιτικού πλουραλισμού, παραδείγματο χάρη, Κομισιόν και το Τσεχικό Υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσαν ένα σχετικό σεμινάριο για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο τον Ιούνιο του 2008. Και εκεί πέρα υπήρχαν υψηλοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της κοινωνίας των ε, πολιτών, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί και ε, δικοί εισηγητές του ΟΗΕ. Εγκρίθηκαν εκεί κοινέ συστάσεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος ε, όσον αφορά παραδείγματος χάρη την ελευθερία έκφρασης, πολέμηση των βασανιστήριων, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη το 2009 είχαμε ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο όπως ξέρετε συνέταξη κομισιόν για τη Μεσογειακή Ένωση και εκεί πέρα προτείνουμε να εξελιχθούν περαιτέρω αυτά τα θέματα. Βεβαίως είναι δύσκολο να βρούμε κοινούς παρανομαστές καθώς γνωρίζουμε την πολιτική πραγματικότητα στην περιοχή αλλά αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για να κλείνουμε τα μάτια στις βασικές δημοκρατικές αρχές και τις κοινές αξίες παρά το στασιμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δραστηριότητες αυτές λόγω βεβαίως τη απόφασης ε, της Αιγυπτιακής Συμπροεδρίας ελπίζουμε ότι το πρόγραμμα εργασίας του 2009 θα διεξαχθεί όπως αποφασίστηκε από τους υπουργούς ε, της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης ε, πέρυσι τον Νοέμβρη στη Μασαλία. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης παρούσης κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με την πολυμερή και με τη διμερή του διάσταση στην Ευρωμεσογειακή Λεκάνη. Πρόκειται για κάτι το οποίο μας εμπνέει στην δράση μας και ποτέ δεν είμαστε αδιάφοροι στο τι συμβαίνει και όσον αφορά τις γενικές αρχές και όσον αφορά τα γεγονότα. Και γνωρίζουμε πως αυτή δεν είναι προσπάθεια της Κομισιόν μόνο, είναι κοινή διοργανική προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντική και για το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοράλ. Το λόγο έχει τώρα ο Γενικός Γραμματέας της ε, πλατφόρμας των μη κυβερνητικών οργανισμών της Euromed. Θα μας, ε, δώσετε, ε, θα μας παρουσιάσετε όλες τις σημαντικές επιτυχίες στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο, κύριε Τουμπιανά αν μπορείτε να μας πείτε σε ποιο μέτρο θα συσταθούν κάποια όργανα ενίσχυσης του ρόλου των μη κυβερνητικών οργανισμών στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας. Κυρία Πρόεδρε, των Προετέρων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε εδώ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε ποιο πλαίσιο οργανώνουμε τις παρεμβάσεις μας. Δηλαδή η πλατφόρμα ε, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε αναγνωριστεί ως ε, θεσμικός εταίρος της Κομισιόν και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων με την υποστήριξη συγκεκριμένα της Κομισιόν που θα ήθελα να ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία. Έστω και αν ε, ως ε, αφετηρία, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας της Βαρκελόνης έχουμε, και αυτός είναι ο ρόλος μας, λιγότερη αισιοδοξία δυστυχώ όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία και της πρόοδου που σημείωσε σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει να πω ότι πολλές φορές αναφέρεται μια χώρα την οποία επισκεφτόμαστε πολύ συχνά. Ε, είναι το Μαρόκο, μια χώρα που δεν μπορεί όμως να είναι το δέντρο το οποίο κρύβει το δάσος ανεξάρτητα από το ζήτημα της διένεξης Ισραήλ και Παλαιστίνης. Και υπάρχουν αρκετές οπισθοχωρήσεις εκεί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όσον αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση. Είναι ένα τελές αποτέλεσμα της διαδικασία της Βαρκελόνης το γεγονός ότι οι πολιτικές των συμφωνιών σύνδεσης ή οι πολιτικές γειτονίες δεν επέτρεψαν, έχω την εντύπωση, να βελτιωθεί με σημαντικό τρόπο η κατάσταση και το γεγονός ότι δίδονται κάποιοι υπολογιστές και λοιπά ή υποβοηθεί το δικαστικό σύστημα ε, είναι καλό αλλά παρόλα αυτά έχει δραματικές επιπτώσεις για τους πολίτες η κατάσταση αυτή. Και το θέμα λοιπόν δεν τίθεται με όρους ποσοτικούς, αλλά κυρίως ποιοτικούς όσον αφορά την εξέλιξη των κανόνων ε, σε σχέση με τη δημοκρατία. Και μιλάμε για εφαρμοσμένους ε, κανόνες ε, σε σχέση με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα βεβαίως. Και αυτό πόσο μάλλον που είμαστε μπροστά σε μια οπισθοχώρηση ε, σε μία μάλλον επιδίνωση της θέσης της κοινωνίας των πολιτών. Οι ακτιβιστές ε, διώκονται, ε, οργανισμοί μη κυβερνητικοί πάβουν να υφίστανται ή εφαρμόζονται έλεγχοι στα κονδύλια υπέρ αυτών των εργανώσεων, συμπεριλαμβάνομαι και αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόκειται για πραγματικά πλήγματα, ε, ε, ακόμα και διώξεις έναντι των ακτιβιστών και ποινές ε, φυλάκισης. Ε, κάποιος αγωνιστής φυλακίστηκε για δύο χρόνια στη Γαλλία επειδή υπερασπίστηκε κάποιον ε, Τινήσιο που ζει στη Γαλλία. και είναι σαφές ότι δεν συμμεριζόμαστε στο επίπεδο αυτό αυτή την κατάσταση και είμαστε λίγο απογοητευμένοι. Και σε αυτή τη συγκυρία βλέπουμε να συστήνεται η Ένωση για τη Μεσόγειο. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό στην αρχή. Ε, μας είχε φανεί πολύ καλός ιονός ε, σε σχέση με τη συνοχή και την ένταξη στη διαδικασία της Βαρκελόνης, στη σχέση με την Κομισιόν ε, και χάρη στις πολύ πλούσιες συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα της Γαλλίας και της Γερμανίας αλλά και άλλων χωρών, η διαδικασία Ένωση για τη Μεσόγειο ενέταξε τη διαδικασία για τη Βαρκελόνη και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ θετικό γιατί υπήρχαν κάποια κεκτημένα στη διαδικασία της Βαρκελόνης και έχουν δρομολογηθεί κάποιες πολιτικές γειτονίες και κάποιες πολιτικές αξιολόγησης ε, των πολιτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Και θεωρούμε ότι η Ένωση για την ε, Μεσόγειο είναι πολύ θετικό είναι πολύ θετικό να ενταχθεί η Ένδονη τη Μεσόγειο σε αυτή τη διαδικασία. Και ε, αλλά πέρα από αυτό έχουμε πολλά ερωτηματικά. Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε μια διαδικασία η οποία αρχικά έχει εξαγγελθεί ότι θα εφαρμόσει πολλά προγράμματα που σχετίζονται με μια βιώσιμη εξέλιξη, έναν σεβασμό του περιβάλλοντος. Ε, προγράμματα στα οποία δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει να επανεξαταστούν ε, τα προγράμματα οικονομικής ε, εξέλιξης αυτών των χωρών, ούτε ώστε να μπορούν να υποφεληθούν από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Και υπάρχει μια διχοτομία δηλαδή από τη μία είναι τα οικονομικά προγράμματα που σχετίζονται με την Ένωση για την Μεσόγειο. Για τα υπόλοιπα το Κοινοβούλιο δεν γνωρίζει πολλά πράγματα και υπογραμμίσαμε ότι η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και οι συγκρούσεις που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές ε, θα πρέπει να συνδεθούν ε, με έναν τρόπο με την Ένωση για την ε, Μεσόγειο. Ε, σήμερα ξέρουμε ότι η διαδικασία έχει παγώσει λόγω της ε, σύραξης ε, Ισραήλ και Παλαιστίνης και σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε τα πάντα έχουν παγώσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε πολλά ερωτηματικά γιατί δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει ποιο, ποια είναι η θέση που έχουν ζήτημα της δημοκρατίας, της διακυβέρνησης και δικαιωμάτων του ανθρώπου εντός του πλαισίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Απριόρι πρόκειται για κάποια κεκτημένα τα οποία θα συνεχίσουν να εκφράζονται μέσω της πολιτικής γειτονίας. Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Ε, πρόκειται για κάποια κεκτημένα της διαδικασίας της Βαρκελόνης τα οποία θα εξελιχθούν εκ παραλίλου με τα οικονομικά και κοινωνικά προγράμματα με ποια μέσα του διαλόγου με τις χώρες εμείς ε, θέτουμε όλα αυτά τα ερωτηματικά. Από την εμφάνιση μιας συμπροεδρίας, η κοινωνία των πολιτών προσέκρουσε σε μια απόρριψη της δικής της συμμετοχής στο εσωτερικό της Ένωσης για τη Μεσογείου, τουλάχιστον σε μια από τις διασκέψεις της όσον αφορά την, ε, σε σχέση με τη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης, όπου η παρουσία της πλατφόρμας που είχε πολύ ενεργό ρόλο στη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης με το δίκτυο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έγινε μια συζήτηση μια ημέρα με αντικείμενο ακριβώς το δικαίωμα συμμετοχής αυτής της πλατφόρμας στη διάσκεψη. Ε, και τελικά αποφασίσαμε ότι στη συνέχεια θα έπρεπε να εξαφανιστούμε εντελώ από τη σκηνή μέχρι να διευκρινιστούν ακριβώς τα δικαιώματά μας και η θέση μας. Εάν ε, ένα τμήμα της εταιρικής ε, ευρωμεσογειακής σχέσης, εποφελούμενο από τη συμπροεδρία, εποφελούμενο από τις νέες δομές της Ένωσης για τη Μεσόγειο, θα μπορέσει, ε, όχι συγγνώμη, θέτει ένα αμφιβόλο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζεται σε πλατιά βάση από την ε, Κομισιόν από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά συνέπεια γιατί πρόκειται εδώ για την κοινωνία των πολιτών της Νοτίου Μεσογείου, όχι της Βορείου Μεσογείου. Εμποδίζεται λοιπόν από την αυτόνομη έκφρασή της η κοινωνία των πολιτών προφανώς οι προοπτικές ε, κάποιων κοινών αξιών και κάποιων κοινών διαβημάτων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία έχω την εντύπωση ότι περιορίζονται σημαντικά. Δεν θα ήθελα εδώ να παίξω την Κασάνδρα όσον αφορά το μέλλον ε, και να προφητεύσω τα χειρότερα. Αυτό το οποίο όμως διαπιστώνω σήμερα είναι ότι από τη μία ήδη υπήρξαν κάποιες εκδηλώσεις απόρριψης απέναντί μας και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι κομισιόν ήταν ε, παρούσες και υποστήριξαν τη δική μας ε, συμμετοχή, όλα αυτά δεχτήκαμε εμείς αυτή την απόρριψη. Κατά δεύτερο λόγο δεν κατανοώ πώς θα εκφραστούν τα ζητήματα αυτά της ε, αξιολόγησης που εκφράζεται μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινωνίας, των συμφωνιών που έχουν συναυθεί των στοχευμένων συμφωνιών που έχουν συναυθεί με συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων πρόοδων ε, και περιλαμβάνοντας και τα προηγούμενα κεκτημένα αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές. Και ε, αν θέλαμε να κάνουμε ένα απολογισμό, ο απολογισμός βεβαίως είναι θετικός και συμμεριζόμαστε την άποψη βάσει της οποίας παρόλα αυτά απομένουν πολλά πράγματα να γίνουν και θα κάνουμε πολλά πράγματα, οφείλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν το παρελθόν και το παρόν έχουμε ένα ερωτηματικό, αλλά όσον αφορά το μέλλον έχουμε ένα διπλό ερωτηματικό. Δηλαδή πώς θα μπορούν να εκφραστούν οι παρεμβάσεις του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων εν γέννη ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρηστή διακυβέρνηση. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Αλλά επίσης μέσω ποιων μηχανισμών η κοινωνία των πολιτών μπορεί πλέον να εκπροσωπηθεί. Και θα έλεγα ότι μια εκπρο... Ε, πρόκειται για μια βεβαίως βέβαιη, εδώ το διακύβουμε, το είναι μια, συγγνώμη, βέβαιη ε, εκπροσώπηση που να μην τίθεται να αμφιβόλω. Γιατί αλλιώς, εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αν δεν είναι εγγυημένη η συμμετοχή μας, δεν θα μπορεί να υπάρξει μια αποτελεσματική συνέχιση των εργασιών. Βεβαίως μπορούμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά με ποιο τρόπο. Και διερωτώ για την, ε, ποια είναι η δομή της συμπροεδρίας ε, που θα μπορούσε να ασκήσει ένα ιονί δικαίωμα βέτο σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή σε σχέση με τη συγκεκριμένη παρουσία ε, μιας, ενός μη κυβερνητικού οργανισμού ή ενός φορέα της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα η Ένωση για την Μεσόγειο να μην περιοριστεί σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα αλλά να αναλάβει πλήρως ε, θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρυσής διακυβέρνησης και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να υπογραμμίζω ότι ναι, είναι πολύ καλό να εφαρμόζονται σημαντικά οικονομικά προγράμματα εάν, εάν αυτό έχει σαν συνέπεια να καταλήγουν σε καταστάσεις ε, διαφθοράς ή να χάνονται, να βυθίζονται μέσα στη διαφθορά τελικά τα προγράμματα αυτά θα είναι εις των κατοίκων και των περιοχών αυτών αλλά εις ολίγων. Ιδού λοιπόν οι ανησυχίες μας, τα προβλήματά μας, οι αγωνίες μας αν θέλετε και ε, ιδού και τα ε, τιματά μας γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραμένει πιστή στις αξίες και στις δεσμεύσεις της, δηλαδή στη σύναψη μιας εταιρικής σχέσης η οποία όμως να μην είναι απογυμνωμένη από βασικές αξίες και αρχές, θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλώς τα πράγματα, την κατάσταση, θα πρέπει να διατυπωθούν κάποιοι όρι, όχι ε, καθέδρας, όχι, όχι να φερθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια ηγεμονική δύναμη, αλλά να θέσει κάποιους όρους, να διατυπώσει κάποιους όρους που να επιτρέπουν μια εξέλιξη της κατάστασης και να δώσει τη θέση που της αρμόζει στην κοινωνία των πολιτών, γιατί η κοινωνία των πολιτών είναι αυτή η οποία πραγματικά επιφορτίζεται με ζητήματα που αφορούν την ε, ισότητα ε, ε, και είναι ένας από τους βασικούς μοχλούς, όπως φάνηκε και στη συνδιάσκεψη της Κωνσταντινούπολης, για την εξέλιξη των κοινωνιών μας εν γέννη. Σας ευχαριστώ για τη θαυμάσια παρέμβαση. Πολλά ερωτήματα θέσατε. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί ορισμένα από τα ερωτήματα του κυρίου Τουμπιάννα μπορείτε να τα απαντήσετε εσείς ως εκπρόσωπος της Επιτροπής ή μπορείτε να αποπειραθείτε. Ε, πώς πιστεύετε ότι θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία, Φερρυπίν. Ο κύριος Μάικλ Έμερσον δημοσίευσε ένα άρθρο για αυτό το θέμα. Θα μας μιλήσει για τους προβληματισμούς του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά θα μιλήσω μετά τους ε, επόμενους ε, ομιλητές. Θα μιλήσω ε, για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ευρία έννοια. Θα μιλήσω για την κοινοβουλευτική δημοκρατία και για τις συγκρούσεις που υπάρχουν στη σχέση τους με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Θα μιλήσω λοιπόν λίγο για αυτά τα τρία θέματα. Καταρχάς θα θέλω να σχολιάσω όμως τα σχόλια που ακούστηκαν για την Ένωση για τη Μεσόγειο, ε, για την ε, Γραμματεία, για τη Συμπροεδρία, για τις ε, Συνόδους Κορυφής. Έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία. Τι, άλλα, τι άλλο όμως έχουμε. Σίγουρα, όπως είπε η κυρία Ναπολιτάνο, έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σε στρατηγικό πολιτικό επίπεδο το θέμα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όμως απέχουν, δεν υπάρχουν με εξαίρεση ε, δύο-τρία έτσι στοιχεία και αναφορές στις ε, επίσημες ανακοινώσεις. Δηλαδή τα προγράμματα αυτά δεν αφορούν τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή, αυτό προκύπτει από την όλη πρωτοβουλία. Ε, από στρατηγική πολιτική άποψη λοιπόν δεν μπορεί να θεωρήσουμε ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο βοηθά τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά καθεαυτά. Το πιο σημαντικό στοιχείο που υπόθηκε είναι ότι η Αιγυπτιακή Συμπροεδρία της Ένωσης για τη Μεσόγειο αποφάσισε να μην συμμετάσχει αυτή τη συνεδρίαση. Τι συμβαίνει στην Αίγυπτο. Θα ήθελα να σας μιλήσω για την, τους αδερφούς μουσουλμάνους. Ο αρχηγός τους ε, έχει συλληφθεί και έχει συρθεί ενώπιον ε, πολιτικού δικαστηρίου για φοβερά αδικήματα. Αυτά τα αστικά δικαστήρια ε, αποφάνθηκαν ότι δεν υπάρχει βάση για αυτή τη δίκη, για αυτές τις διώξεις. Φαντάζομαι το επόμενο βήμα είναι να πάει το θέμα αυτό σε στατιωτικά δικαστηρία. Αυτό είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Καταφανής παραβίαση. Νομίζω ότι πέρασε χωρίς να αναφερθεί καθόλου. Δεν ξέρω τι διπλωματικά διαβήματα έκανε η Κομισιόν και η αντιπροσωπεία των κρατών μελών, αλλά αν υπήρξαν αυτά διαβήματα ήταν τόσο ήπια που πέρασαν απαρατήρητα. Ε, δεν είναι καλές αυτές οι επιδόσεις, έτσι. Τώρα από την πλευρά της δημοκρατίας. Το θέμα είναι πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα συνδεθεί με αντιπάλους που αγωνίζονται για να αποκτήσουν και αυτοί τι βήμα στην πολιτική σκηνή. Παραδείγματο χάρη, τα Ισλαμικά κόμματα συχνά αποκλείονται ή η παρουσία του είναι εντελώ συμβολική. Δύο από του συναδέλφου σα, ε, Πρόεδρε, δημοσίευσαν ένα θαυμάσιο βιβλίο πέρυσι που λέγεται «Η αναζήτηση για τη δημοκρατία». Ε, ταξίδι προς τη δημοκρατία των ε, μουσουλμάνων γειτόνων μας γίνεται μια αποτίμηση του πώς τα μετριοπαθή Ισλαμικά κόμματα ουσιαστικά αποκλείονται. Για να, εν πάση περιπτώσει αποθαρρύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Τώρα, αυτό συνδέεται με την ε, μεταχείριση της Χαμάς, που την αντιμετωπίζουμε ως τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν δύο στοιχεία σε αυτό. Καταρχάς, είναι σαφές σε όλο τον γραφικό κόσμο ότι η συνεχής άρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλήσει, να συνομιλήσει με τη Χαμάς και το γεγονός ότι την κρατάει τη Χαμάς στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων οδήγησε σε παράπονα α, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διπλά πρότυπα, διπλά μέτρα και σταθμά. Τώρα, για την ίδια τη Χαμάς Συζήτησα με τον πρεσβευτή ενός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πρόσφατα και του είπα μήπως είναι καιρός να αρχίσουμε να συνομιλούμε με τη Χαμάς μια και είναι μέρος, τμήμα όλων αυτών των δραματικών ε, ε, τεκτενόμενων. Ακόμη και η Ρωσία μιλάει με τη Χαμάς. Ε, αυτός τι μου απάντησε μιλήσαμε με την Νορβηγία. Τελεία. Αυτή η σχέση, μάλλον η έλλειψη σχέση με τη Χαμάς, είναι τμήμα του προβλήματος και δημιουργεί τεταμένες καταστάσεις. Όχι μόνο με, την, με το θέμα της Παλαιστίνης, αλλά και με το θέμα της Αχέλ που ακούστηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει διαπραγματεύσεις για συμφωνίες σύνδεση με το Μαρόκο και το Ισραήλ. Ε, και το Ισραήλ, συγγνώμη. Ε, σταματήσαμε τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Δεν ξέρω αν είμαστε ακόμη σε φάση αναστολής ή αν ξανασυνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις σοβαρότατα προβλήματα. Και δυστυχώς η Ισραηλινή Δημοκρατία με την ε, κομματική δομή που έχει, θα έχουμε σήμερα τα αποτελέσματα των εκλογών. Νομίζω ότι θα δούμε ότι θα υπάρξει μια κίνηση προς τα δεξιά. Η ακροδεξιά του Ισραήλ είναι πραγματικά ριζοσπαστική και δίνει μηδενική προοπτική για ειρήνη στην ε, περιοχή. Φυσικά η κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει την ε, επέκταση των ε, οικισμών και με άλλες παραβιάσεις των νομικών της δεσμεύσεων. Αυτό είναι το πλαίσιο. Εκεί μέσα αναπτύσσονται οι ριζοσπαστικές τάσεις στα παλαιστινιακά εδάφη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει απλώς δηλώσεις για, για να αποδοκιμάσει το ένα και το άλλο. Αλλά αυτές οι δηλώσεις οδηγούν σε στοιχεία τα οποία είναι καθαρά συμβολικά και δεν, έχουν, και δεν επηρεάζουν καθόλου την, ε, την κατάσταση. Τώρα, η μαροκινή περίπτωση είναι λιγότερο χτυπητή. Έχουμε τεράστιους, τεράστιο αριθμό προσφύγων ε, στα δυτικά που ζουν σε φρικτές καταστάσεις ε, και η μαροκινή κυβέρνηση που είναι ο κατακτητής, μπλοκάρει τη διαδικασία στον ΟΗΕ που ζητάει να γίνει δημοψήφισμα για να επιληθεί η κατάσταση. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει τίποτα. Ένα τελευταίο ζωφερό ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Αυτή η αδύναμη διάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι εντελώς μηδενική. Βέβαια, η Κομισιόν με μεγάλη προσοχή και σχολαστικότητα περιέγραψε τις διαδικασίες που προσπαθεί να προωθήσει η Κομισιόν στα πλαίσια ιδίως της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Εγώ ως πρώην υπάλληλος της Κομισιόν καταλαβαίνω τους πολιτικούς περιορισμούς μέσα στους οποίους κινείται η Κομισιόν και με τους οποίους προσπαθεί να δώσει διάσταση στη, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά από στρατηγικής απόψεως πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η δραστηριότητα είναι για τους τύπους, είναι συμβολική. Και όπως είπε και η κυρία Ναπολιτάνο, δεν έχουμε καθόλου αυτά αποτελέσματα. Τώρα, το αν είμαστε πραγματικά προς το, τίνουμε στο μηδέν, αν είμαστε στο μηδέν, ή αν όχι έχω να σας πω ότι όλα αυτά τα στοιχεία οδηγούν στην αύξηση του ριζοσπαστισμού στον αραβικό μεσογειακό κόσμο, ε, στην Τουρκία και αλλού. Υπάρχει μια σχετική μελέτη πρόσφατη δεν μπορώ να πω ότι τα στοιχεία της μελέτης είναι καθαρά επιστημονικά και αδιαμφισβήτητα, αλλά υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα σε αυτή τη μελέτη ότι η αδύναμη αυτή πολιτική συνομιλίας με το δημοκρατικό Ισλάμ και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικά βοηθάει τους ριζοσπάστες, τα Ισλαμικά κόμματα που είναι ακραία και σίγουρα αν αυτό δεν είναι μηδενική προσπάθεια, τουλάχιστον μη σας πω ότι δεν είναι αρκετή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δώσουμε το λόγο στα μέλη μας. Ο κύριος Σουμπιότς. Α, Ρεϊμόν ε, ε, θα πρέπει να πάρεις το λόγο γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ε, κυρία Πρόεδρε, θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί πραγματικά καθυστέρησα να φτάσω, γιατί είχε τεράστιο μποτιλιάρισμα ε, και είχε κοπεί η συγκοινωνία στην ε, Λεφόρο και δεν μπόρεσα να ακούσω όλες τις παρεμβάσεις. Γι' αυτό θα αναφερθώ σε αυτό που άκουσα συγκεκριμένα στην παρέμβαση του κυρίου Τουμπιάνα και του κυρίου Μάικλ Έμερσον. Έχω την εντύπωση ότι συνεχίζουν ε, μία γραμμή σκέψης σε σχέση με τις ανησυχίες που αισθανόμαστε όσον αφορά τη γενική κατάσταση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μεσόγειο από τη μία, της Ένωσης για τη Μεσόγειο, ε, διαδικασία που έχει παγώσει αυτή τη στιγμή, συνεπία ακριβώς της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης και τα όσα συνέβησαν στη Γάζα. Από την άλλη υπάρχει μια ανησυχία την οποία εγώ θα νόμιζα στο πλαίσιο μια συζήτηση που είχαμε με την Γαλλική Προεδρία ε, μια υπερβολή της Real Politik ε, στο επίπεδο των ευρωμασογειακών σχέσεων. Δηλαδή ένα όραμα μέσω του οποίου ο θεμελιώδης στόχος, δηλαδή η εξέλιξη των μεγάλων ε, προγραμμάτων στην περιοχή αυτή, οικονομικής εμβέλειας, δημιουργία υποδομών κλπ. κλπ. Αλλά βεβαίως αν συγκρίνουμε ε, ε, τις εξαγγελίες αυτές με τα όσα συνέβησαν υπάρχει μια δυσαναλογία. Ε, βέβαια υπάρχει μια σύγχυση στην κοινή γνώμη όσον αφορά αυτές τις εξελίξεις, αλλά σε όλους τους ε, τομείς, ε, στην πολιτική, στους μη κυβερνητικού φορείς, η διάσταση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η υπεράσπιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μοιάζει να έχει οπισθοχωρήσει σε σχέση ε, με την ε, με, την, ε, με τις πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί. και δεν είναι πολύ ξεκάθαρη εξελίξη στο πλαίσιο τη διαδικασία τη Βαρκελόνη. Συνεπώ, κατά πρώτο λόγο θα ήθελα να πω και δεν μιλώ προσωπικά, αλλά εκπροσωπώ όσους ε, παρακολουθούμε τα θέματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν μια πιστοχώρηση. Βεβαίως το να θλιβόμαστε για αυτή την κατάσταση αυτό δεν είναι ιδιαίτερο ε, χρήσιμο. Ε, μας καθιστά μόνο μελαγχολικούς. Ε, το ζήτημα είναι πώς θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Η διαδικασία συγκρότησης της Ένωσης για τη Μεσόγειο είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη, όπως επεσήμενε ο κύριος του και από μια περίοδο σχετικής σύγχυσης έχει εξελιχθεί σε μια φάση ένταξης της διαδικασίας της ε, Βαρκελόνης και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση τώρα ε, που βεβαίως αν βγούμε από την παρούσα στασιμότητα θα περάσουμε σε μια φάση εφαρμογής. Ε, και θα πρέπει να ενταχθούμε σε αυτή τη νέα θεσμική πραγματικότητα για να ενισχύσουμε περισσότερο αυτή τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε πώς και με ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις τα επόμενα χρόνια. Γιατί από τη μία έχουμε την παρούσα στασιμότητα, το πάγωμα της διαδικασίας, την παρούσα συγκυρία. Δεν γνωρίζουμε εάν οι αντιπαραθέσεις, η σύγκρουση στην Εγγύης Ανατολή θα γνωρίσει μια διακοπή, θα σταματήσει μάλλον ή θα υπάρξουν νέες επιθέσεις. Ε, κατά την άποψή μου ε, πρόκειται για μια δαμόκλια, ε, υπάρχει εδώ μια δαμόκλια σπάθη που κατά την άποψή μου είναι ευνοϊκή, είναι η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Και ο κίνδυνος μίας παρέμβασης εκ μέρους του Ισραήλ σε σχέση με τις ε, πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε μια τρομακτική έκρηξη σε όλη την περιοχή, στο Λίβανο, στη Γάζα ε, και σε όλες τις γειτονικές ε, χώρες την Ορδανία κλπ. Και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση τόσο μεγάλων ανησυχιών και φόβων που κατά πάσα πιθανότητα, και μιλάμε τώρα για τις επιπτώσεις που θα έχει στην Ένωση για τη Μεσόγειο, ούτως ώστε να υπάρξει μια, ένας αυτοπεριορισμός. Υπάρχει ένας, ένα άλλο στοιχείο που εγώ θεωρώ ανησυχητικό. Είναι ότι οι πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου νομίζω υλοποιούν ε, τη φράση του Ναπολέοντα ε, κανείς ε, αναλαμβάνει μια δέσμευση και στη συνέχεια περιμένει να δει τι θα γίνει. On s'engage puis και υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, ενισχύσουμε την αισιοδοξία της ε, βούλησης για να μην αναστείλει τις προσπάθειές μας η απεσιοδοξία της λογικής. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις στο τέλος αυτής της θητείας ούτως ώστε να υπάρξει ένα στρατηγικό όραμα ανάπτυξης, εξέλιξης στην περιοχή αυτή, στη Μεσόγειο, που να βασίζεται όχι μόνο στην ελεύθερες συναλλαγές και στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στον εκδημοκρατισμό και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό με ένα μεγαλύτερο δυναμισμό από ό,τι έγινε στο παρελθόν. Κατά δεύτερο λόγο, η αντίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η πρόθεση μάλλον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την υποεπιτροπή αυτή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι μια ε, επιπλέον διάσταση στα οικονομικά προγράμματα και θα πρέπει να εμπνέει τις πρωτοβουλίες ε, των ε, πολιτικών που θέλουν να κάνουν αυτή τη διάκριση, αυτό τον διαχωρισμό. Εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε, να προθίσουμε ένα υπόδειγμα βάσει του οποίου τα οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτιστικά και ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι ο βασικός άξονας των δράσεών μας. Έλαβα γνώση των όσων ελέγχθησαν εδώ ε, και για το βιβλίο σχετικά με την ριζοσπαστικοποίηση του Ισλάμ στη Μεσόγειο, ε, το βιβλίο που έγραψαν από κοινού η Βίρσμα και Λάγκεντικ. Νομίζω ότι θα πρέπει, όπως λένε στην Ισπανία, να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε αντίθετα στο ρεύμα, όσο και αν τα ρεύματα αυτά είναι πολύ απειλητικά και απειλούν να μας παρασύρουν. Ευχαριστούμε πολύ. Πασκαλίνα, θέλεις να ξαναπάρεις το λόγο. Όχι, μου φαίνεται πως ε, υπάρχει εδώ πέρα μια βασική συμφωνία σε αυτά τα οποία λέγονται και εγώ θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε χρειάζεται ένα όραμα το οποίο δεν θα καλύπτει μόνο τις οικονομικές πτυχές λείπουν άλλες πτυχές που δεν έχουν νομίζω τονιστεί αρκετά γιατί αυτή η ρεάλ πολιτική επικρατεί στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. για το ζήτημα της μετανάστευσης και η διαχείριση αυτών των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες... Όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Κύπρος, που είναι οι χώρες που βρίσκονται στην πρωτοκαθεδρία αθνοσχέσεων. Συχνά είναι οι χώρες που έχουν, επειδή έχουν πολλά προβλήματα λαθρομετανάστευσης, αντιδρούν ζητώντας την εταιρική σχέση με τις μεσογειακές χώρες να η σχέση αυτή να διέπεται από μια προσπάθεια καταστολής της λαθρομετανάστευσης αδιαφορώντας πλήρως για τις επιπτώσεις αυτής της καταστολής. Καταλαβαίνετε ότι όταν γίνεται, γίνονται επιχειρήσεις επαναπροώθηση στα σύνορα χωρίς να εξασφαλίσουμε ότι τα άτομα αυτά αντιμετωπίζονται με σεβασμό και σεβόμαστε την, ε, τη ζωή τους και τα δικαιώματά τους, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πώς να ισχυριστούμε μετά ότι είμαστε μεταξύ αυτών ε, που προωθούν στις χώρες αυτές τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στην όλη πρόπτικη. Εάν δεν αλλάξει η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο θέμα αυτό, γιατί να σας πω κάτι, δεν θα έχουμε καν και το δικαίωμα, αν θέλετε, να οδηγήσουμε προς τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτή την εταιρική σχέση. Συμφωνώ ότι δουλεύουμε σε δύσκολες συνθήκες. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι και τα κινήματα των, ευρωπαϊκών κοινωνιών, της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια σύνδεσης με την κοινωνία των πολιτών των νοτίων χωρών της Μεσογείου. Έχουμε τεράστια προβλήματα και στην Ευρώπη, μην το ξεχνάμε. Εμείς δεν είμαστε στο απειρόβλητο. Θα ήθελα να αναφέρω την περίπτωση της Ιταλίας, για να μην μιλάω άσχημα για άλλες χώρες. Στη χώρα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανείς την Ιταλική ηθαγένεια, για να μην πω σχεδόν αδύνατο έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Ακόμη και τα παιδιά τα οποία γεννιούνται στην Ιταλία δεν έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν ποτέ την Ιταλική υπηκότητα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι περίπου ένα 10% και αυτή η τάση είναι όλο και αυξανόμενη θα φτάσει στο 20% πολιτών, γιατί εγώ πώς να τους ονομάσω αλλιώς. Πολίτες πρέπει να τους ονομάσω. Δηλαδή υπάρχουν πολίτες που δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. Εμείς στο σύνταγμά μας του 48 πολεμήσαμε για να δώσουμε το καθολικό δικαίωμα ψηφοφορίας σε, ανθρω... σε γυναίκες, άνδρες, φτωχούς, πλούσιους. Σήμερα όμως Έχουμε μια κοινωνία όπου ένα τμήμα δεν έχει πολιτικά δικαιώματα, δεν συμμετέχει σε, αυτή την, σε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε δηλαδή, ε, αντιμετωπίζουμε σοβαρό κίνδυνο αντιστροφής ε, της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό δεν αισθάνομαι ότι είμαι σε θέση ως Ευρωπαία να υποδείξω με το δάκτυλο στο, στους Αιγύπτιους, στους Μαροκινούς τι πρέπει να κάνουν. Πιστεύω πραγματικά πολύ στην εταιρική σχέση. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κίνδυνοι οπισθοχώρησης και στις δικές μας κοινωνίες. Γι' αυτό η ενδυνάμωση μια στρατηγική σχέση από πλευράς κυβερνήσεων, ε, κοινοβουλίων και κοινωνία των πολιτών είναι ο μόνος τρόπος για να προλάβουμε τις ε, επιπλοκές. Σε όλα αυτά τώρα θα ήθελα να βάλω και ένα στοιχείο ελπίδα σε σχέση με αυτά που είπε ο Ιράν, ε, ο, ο Ρεϊμούν για το Ιράν. Μην ξεχνάμε ότι τον ε, Ιούνιο θα γίνουν οι εκλογές. Ο Κατάμι θα κατέβει στις εκλογές και ελπίζουμε ότι εκείνο το τμήμα της κοινωνίας του Ιράν που δεν ψήφισε και επέτρεψε τον Αχμαντινετζάν να νικήσει, αυτή τη φορά θα συμμετάσχει στις εκλογές και επομένως ίσως κάτι αλλάξει στις σχέσεις μας με το Ιράν. Ευχαριστώ. Euh, ε, λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι ε, αν κάποιες ερωτήσεις δεν τεθούν ανοιχτά στο τραπέζι θα έχουμε μεγάλη, να αντιμετωπίσουμε μεγάλη δυσκολία στο να εκπονήσουμε κάποιους θεσμούς που να αγγιούνται τη συμμετοχή, να τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη δικασία αυτή και ε, να υπάρχουν και πολυμερείς συμφωνίες. Να υπάρξουν δηλαδή, κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, Βεβαίω, ε, κάθε φορά αναφέρεται το παράδειγμα του Μαρόκου. Εγώ όμω θα ήθελα να αναφέρω την, ε, την Ισία. Αυτή η μικρή χώρα που δεν έχει πετρέλαιο και με την οποία συνήφθη η πρώτη συμφωνία σύνδεση στην περιοχή αυτή είναι αδύνατον μέχρι στιγμής να υπάρξει μια σωστή, ένα σωστός στρατηγικής ή πολιτικής που να φέρνει κάποια από τα αποτελέσματα. Αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς. Μια υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από ένα μήνα ε, κλείστηκε στη λάσπη από τον τύπο της ε, κυβέρνησης ε, το, τα γραφεία λατήθηκαν, ο εξοπλισμός εκλάπη κλπ. Ή ένας εκπρόσωπος ε, κάποιων ε, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Μαγκρέμπ ε, επίσης δέχτηκε πολλές ε, επιθέσεις. Ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Συνεπώς το μόνο θέμα που μπορούμε να θέσουμε αν κατά πόσο στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο θα εξεύρουμε τα μέσα μιας νέας, ενός νέου δυναμισμού και αποτελεσματικότητας για να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί έτσι τίθεται το θέμα, έτσι θα πρέπει να τίθεται το θέμα με αυτούς τους όρους. Εγώ δεν ξέρω πώς μπορούμε να μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα με ορισμένε ε, από τις χώρες αυτή τη περιοχή. Εάν δεν μπορούμε σήμερα να υποστηρίξουμε τη διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης ε, διεθνούς έρευνας σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στη Γάζα ε, κατά τη διάρκεια των τριών αυτών εβδομάδων, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες να συνεχίσουμε να έχουμε έναν σοβαρό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί η δική μας αξιοπιστία θα κυλιδωθεί εάν δεν γίνει, γίνουν κάποιες, κάποια σοβαρή εργασία σε σχέση με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με εγκλήματα πολέμου όλες οι συζητήσεις που γίνονται με τους ε, εταίρους μας της ε, Νοτίας Μεσογείου ε, μας παραπέμπουν στη συζήτηση για την οδηγία τις επιστροφές. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τις μεταφορές προσώπων τα οποία τελικά βασανίζονται στα κέντρα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο να συζητούμε για βασανιστήρια ανθρώπων σε κάποιες χώρες, ε, ανθρώπων που έχουν ε, μεταφερθεί στα κέντρα αυτά με τη δική μας συνδρομή. Το να κερδίσουμε εδώ, σε αυτό το, στο πλαίσιο αυτού του διακυβεύματος είναι πραγματικά θεμελιώδες. Ε, είναι ένα θέμα που τίθεται στο επίπεδο του Συμβουλίου. Θα πρέπει να διατυπώσουμε τους όρους που θα μας επιτρέψουν να εξέλθουμε τροποτινά από την εμφανή μας αδυναμία να προχωρήσουμε παρά τους σοβαρούς αυτούς μηχανισμούς που έχουν πράγματι συσταθεί και θα συζητήσουμε, περνώντα στο δεύτερο σημείο τη ημερήσια διάταξη, για το γεγονό ότι η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, για παράδειγμα τη βοήθεια μηχανισμών ε, όπω είναι οι συμφωνίε του Κοτονού που σε περίπτωση παραβίασης ε, θα πρέπει να γίνει σύντηση με την λόγο χώρα ε, και να ληφθούν κάποια περιοριστικά μέτρα, τέλος πάντων να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα αναστολή ε, του διαλόγου σε, κάποια, σε κάποιες περιπτώσεις. Ε, θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη συνείδηση όσον αφορά την ισορροπική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο επίπεδο του Συμβουλίου θα πρέπει να επισημάνουμε, να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ατέλειες, τεράστιες δυσκολίες στο επίπεδο της χάραξης μιας στρατηγικής. Η Ένωση για τη Μεσόγειο αρχικά ήθελε να εξετάσει μόνο τα σημαντικά προβλήματα που δυσχεράνουν την εξέλιξη της διαδικασίας. Όπως για παράδειγμα είναι οι δυσκολία στην προχωρή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Α, συγγνώμη, όπως είναι τα μεγάλα περιφερειακά προγράμματα, βάζοντας κάπως στην άκρη την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τα τρία τέταρτα του χρόνου που, στο Παρίσι ασχοληθήκαμε με τη διαπραγμάτευση της παραγράφου για την ε, Μέση Ανατολή, κάτι το οποίο δεν θέλαμε να συζητήσουμε όμως αρχικά. Και σήμερα η Ένωση για την Μεσόγειο ίσως έχει την ε, ευκαιρία να οικοδομήσει μια νέα αξιοπιστία αποβαίνοντας χρήσιμη ακριβώς στο πλαίσιο της σύγκρουσης της Γάζα. Αυτό θα έπρεπε να συμβεί. Αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο και τα πάντα έχουν παγώσει. Και είμαστε εντελώ ανίσχυροι. Ε, δεν ξέρω πώ θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι που να είναι πραγματικά παραγωγικό και αποτελεσματικό. Υπάρχουν άλλοι βουλευτέ. Όχι. Που να θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στου προσκεκλημένους μα, ξεκινώντα από τον κύριο Δεμοράλ. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για αυτή την τελευταία σας παρέμβαση που κατά κάποιον τρόπο έτσι θέτει το ερώτημα με τους όρους που πρέπει. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που απευθύνθηκαν προς την Κομισιόν ως θεσμικό όργανο. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η θέση της δημοκρατίας και της κυβέρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Μεσογειακή Ένωση. Και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία σε αυτό το πλαίσιο. Οφείλω να πω πως η Μεσογειακή Ένωση έχει στόχους, αρχές, γνωστούς. Έχουμε θεσμικά οργάνα που έχουν οριστεί τα θεσμικά όργανα από μόνα τους είναι ουδέτερα. Απλά προσπαθούν να εγγυηθούν ε, έτσι, μια εμπλοκή στη διαδικασία. Έχουμε έργα, έργα που δεν συμπεριλαμβάνουν στοιχεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, όπως ακούστηκε, και έχουμε λίγους μηχανισμούς. Γιατί όσον αφορά τους μηχανισμούς, αυτό το οποίο έχουμε κυρίως είναι μηχανισμοί διαλόγου συναντήσεις αξιωματούχων, υπουργών που υιοθετούνται προγράμματα τεχνικά κυρίως καμιά φορά και κάτι άλλο το πρόβλημα που έχουμε είναι βεβαίως πως ε, τους γείτονες δεν τους διαλέγει κανείς και η δυνατότητά μας έτσι να τους κάνουμε να συμπεριφερθούν σωστά περιορίζεται από το γεγονός ότι είναι κυρίαρχα κράτη. Δεν το μεταγιώνουμε αυτό. Σωστά είπατε πως αυτοί τις οποίες μπορούμε να επηρεάσουμε είναι αυτοί που θέλουν να γίνουν μέλη. Εκεί ένας τρόπος πίεσης ε, και μπορούμε να βάλουμε όρους και να αποδεκτούς. Αν δεν υπάρχει αυτό, τα ε, βλέπετε τα αποτελέσματα σε πολυμερή πλαίσια όπως αυτό της Μεσογειακής Ένωσης όπου παρά την θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθηθεί η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. και δεν θα πρέπει να βάλει κανείς γι' αυτό, έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. Αυτά τα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό δεν ισχύει τόσο για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, για την οποία είπα πως κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένη, πιο χρήσιμη. Στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία και εμείς ε, και οι εταίροι μας θα με κάποια πράγματα ο ένας από τον άλλον. Και το γεγονός πως υπάρχουν στόχοι, φιλοδοξίες, μας επιτρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Υπάρχει ο ίδιος βαθμός προόδου παντού. Όχι. Σαφώς. Και το γεγονός ότι αναφέρουμε το Μαρόκο απλά το κάνουμε για να δείξουμε πως υπάρχει πρόοδος κάπου. Αλλού όχι. Δεν είναι θέμα διπλών μέτρων και σταθμών, τα μέτρα είναι ίδια, η δυνατότητα πρόοδου δεν είναι ίδια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Επίσης ετέθη το ερώτημα του εάν μπορούμε να έχουμε εγγυήσει για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, π.χ. σε εκδηλώσεις όπου έχει υπάρχει μια απόρριψη. Δεν υπάρχουν εγγυήσει. Δεν υπάρχει ένας μηχανισμός. Πλην του ότι γίνεται μια αναφορά συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, στην διακήρυξη των Παρισίων και σε προηγούμενες διακήρυξεις διαδικασίας της Βαρκελόνης. Τι γίνεται τώρα εάν υπάρχει κάποιος αποκλεισμός. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το βάρος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων έτσι ώστε να μην αγνοούνται οι ανησυχίες μας. Και σε κάποιες περιπτώσεις μπορέσαμε να επιτρέψουμε στην κοινωνία των πολιτών είτε να λάβει μέρος, είτε να κάνουμε ζήτημα τιμή συμμετοχή. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Στην περίπτωση αυτή, αυτό ήταν κάτι που το ήθελε η Συμπροεδρία. Η συμπροεδρία εφόσον ε, μας επιτρέπει την εμπλοκή είναι κάτι το θετικό και το ξέραμε γιατί υπήρχε ένα κενό γιατί όλοι ήθελαν να είναι πιο ισορροπημένη η διαδικασία. Το πρόβλημα είναι πως μόλις γίνει κάτι τέτοιο υπάρχουν και συνέπειες. Και πρέπει αυτές τις συνέπειες ε, να τις αναγνωρίσουμε. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν που εμπλεκόταν πολύ στενά με τη διαδικασία δεν συνδέεται πλέον τόσο στενά ακριβώς γιατί υπάρχει συμπροεδρία. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Να θυμάστε. Ε, τώρα αν αυτό το θεωρείτε, οψοδρόμηση είναι. Αλλά αν θεωρήσουμε πως υπάρχει εμπλοκή των εταίρων μας από την άλλη όχθη της Μεσογείου δεν είναι. Βεβαίως γνωρίζουμε κάποιους κινδύνους. Αλλά σας διαβεβαιώνουμε πως δεν θα υπάρξει οπισθοχώρηση. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα βέτο για το ποια προγράμματα και χρηματοδότηση έχουμε στη διαδικασία αυτή. Γεγονό είναι πως τώρα υπάρχουν νέοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όποια χρηματοδότηση και προγράμματα είχαμε πριν, ε, εξακολουθούμε να τα έχουμε. Δεν έχει διαγραφεί τίποτα, ούτε και πρόκειται. Θα συνεχίσει αυτή η διαδικασία και δεν θα αποδεχτούμε το δικαίωμα του ΒΕΤΟ. Είναι προνόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπεύουμε να συνεχίζουμε να το έχουμε. Που δεν με ανησυχείτε γι' αυτό. Τώρα αναφέρθηκαν οι όροι και το πώς θα έχουμε κάποιες αποτελεσματικές προϋποθέσεις. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα και πώς θα λειτουργήσει. Εάν σπρώξουμε βεβαίω στα άκρα αυτή την ιδέα της ε, ισχύω ε, όσον αφορά την πρόθεση των αξιών μας φτάνουμε στο Ιράκ. Στην άλλη άκρη δεν έχουμε σχέσεις με τους εταίρους μας, με τους γειτονές μας εδώ πέρα. Μπορείτε να τους δείτε εταίρους ή όχι. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε τις σχέσεις που χρειαζόμαστε, γιατί βεβαίως η γειτονία είναι πολύ περισσότερα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την πραγματική σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών. Που θα μας ε, επιτρέψει να ασχοληθούμε με ζητήματα πολύ σημαντικά όπως το οικονομικό χάσματος, το ζήτημα της μετανάστευσης, που σωστά αναφέρατε, και το γεγονός ότι μπορούμε να επηρεάσουμε το, τις κυβερνήσεις αυτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό γίνεται μέσω του διαλόγου, μέσω των κινήτρων, μέσω της αναφοράς σε πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι στο πνεύμα της εταιρικής σχέσης. Τώρα, είναι κάτι τέτοιο αδύναμο, εντάξει, μπορεί να ρωτηθεί κανείς αν μπορεί να είναι πιο δημόσια τα πράγματα, να έχουμε πιο ισχύρη γλώσσα να συνοδεύεται από κάποια μέτρα. Προσπαθούμε να τα εξετάζουμε όλα αυτά τα πράγματα σε σχέση με τους γειτονές μας. Θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια όρια βέβαια στο τι μπορούμε να κάνουμε. Εκτός αν θέμε να, να είμαστε μόνοι μας βεβαίως. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Δεν λέω βεβαίω πως αυτά τα οποία κάνουμε είναι τέλεια. Δεν είπα πως ε, τα όλα είναι εντάξει. Είπα πως η εξολόγησή μας δείχνει πως έχει γίνει κάποια πρόοδος αλλά δεν αρκεί ας είμαστε ρεαλιστές. Σε κάποιες περιπτώσεις σημειώνεται πρόοδος. Όπως το Μαρόκο, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. αλλού δεν έχουμε πρόοδο. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, πάμε και προς τα πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση να κάνουμε. Πρέπει να κινούμαστε στα όρια που, που έχουμε, που υπάρχουν. συγκεκριμένα τώρα για κάποια πράγματα που ακούστηκαν. Πράγματι υπάρχουν συγκρούσεις και οι συγκρούσεις αυτές επηρεάζουν το πώς εργαζόμαστε. Το Παλαιστινιακό υπήρχε όταν ξεκίνησε η διαδικασία της Βαρκελόνης και όριζε τα όρια αυτής της διαδικασίας και το ίδιο σήμερα. Η εμπλοκή των άλλων κρατών το κάνει ακόμη πιο επίγον αυτό το ζήτημα. Επίσης, η δυνατότητα περιφερειακής ολοκλήρωσης στο Μαγκρέπ, Πώ να το αγνοήσουμε. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Θα θέλαμε να υπάρχει δυνατότητα ολοκληρωμένων σχέσεων, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Μακάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έλεγε πως έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε αυτές τις συγκρούσεις, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό το οποίο λέω είναι πως προσπαθούμε να είμαστε ταπεινοί, ρεαλιστές και να κινηθούμε προς τα μπρος. Αλλά δε, βεβαίως πάντα ισχύουν μεύσεις μας, τις αρχές μας και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοράλ. Ο κύριος Τουμπιανά έχει το λόγο τώρα. Θα κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. σε σχέση με το θέμα της διατύπωσης συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Θα ήθελα να πω το εξή. Βρίσκω κάπως απελπιστικό το γεγονός ότι η συζήτηση κάθε φορά ε, γίνεται με όρους του πώς ε, μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα ατομικό όπλο ή έχω τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω ένα ατομικό όπλο. Έτσι ακούγεται. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περάσουμε από τον κριτικό διάλογο ή τη διατύπωση κάποιων όρων στην ατιμορρησία. Δηλαδή να δώσει κανείς πολιτικά την αίσθηση σε ένα κράτος ότι εν πάση περιπτώσει θα βρίσκεται σε καθεστώς ατιμορρησίας. Και παίρνω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έζησε ε, έστειλε μία επιδότηση στο Σύνδεσμο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τινησίας και η επιδότηση αυτή παρέμεινε στην τράπεζα της Τινησίας και δεν ε, δόθηκε ποτέ και χρειάστηκε να γίνει αγώνας ούτως ώστε να επιστραφεί αυτή η επιδότηση για να πάβει να πλουτίζει την Εθνική Τράπεζα της Τινησίας. Αυτόν ναι, εμέν είναι μία μικρή λεπτομέρεια αλλά από την πλευρά των αρχών της Τινησίας ε, θεωρήθηκε σαν μία μορφή ατιμορρησίας. Έτσι έγινε έτσι προσελήφθη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ονειροπόλοι. Ε, δεν μπορούμε να καθίσουμε και από ε, ένα τραπέζι και να πούμε ε, θα κάνεις αυτό ή το άλλο. Ε, ή να στέλνουμε, γιατί μπορούμε τελεσίγραφα, αλλά μεταξύ αυτού και της αδυναμίας όχι να ασκήσουμε πίεση, αλλά να χορηγήσουμε, αλλά να μην δώσουμε την αίσθηση ότι θα υπάρχει πλήρης ατιμορρησία, ζητώντας μια ευθύνη εκ μέρους εκείνων που πραγματικά θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις συγκεκριμένες πράξεις. Δεν αγνώ τη δυσκολία που υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κομισιών κλπ. Και, και Συμβουλίου Υπουργών και των ε, συμφερόντων της κάθε χώρας μέλους σε ένα τομέα όπου η Ευρώπη από πολιτική άποψη παραμένει αδύναμη. Αν θέλουμε όμως να είμαστε συνεπείς ε, ως προς τις αξίες μας, αυτό πώς θα γίνει μόνο να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας. Και το τελευταίο που θέλω να πω. Θέλω να πω εμφατικά ότι Κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών και βουλευτικών εκλογών που έγιναν στα κατεχόμενα εδάφη. Ήδη μετά τις βουλευτικές εκλογές που έφεραν τη Χαμά στην πρώτη θέση Νομίζω ότι μπορώ να πω χωρίς να κάνω λάθος ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές παρόντες εκεί ζήτησαν από τις κυβερνήσεις τους να ξεκινήσει διάλογος ε, με τη Χαμάς και με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Δεν μπορούμε να πούμε στην λαό ψηφίστε. Μπράβο σας. Καταφέρατε να κάνετε εκλογές μέσα σε καθεστώς ε, κατοχής ε, ήταν δημοκρατικές, αλλά ε, δεν τα καταφέρατε όσο καλά θα θέλαμε, γιατί δεν ψήφισατε το σωστό κόμμα. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει να διοργανώσουμε μία ε, ερευνητική επιτροπή για να δει τι έγινε αυτές τις εβδομάδες. Από την άλλη, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η δημοκρατία ε, έχει, γεωμετρι... μεταβλητή γεωμετρία. Και με αυτόν τον τρόπο δεν επιλύονται οι συγκρούσεις. Όλα αυτά αντανακλώνται σε εμά στην κοινωνία των πολιτών. Από τη Γάζα και μετά τα τεκτενόμενα της Γάζας και μετά ποτέ δεν είχαμε... Ε, έχει αυξηθεί τόσο πολύ ένταση που δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ πριν. Δεν μιλάμε καν για διμερείς σχέσεις. Μετά τη Γάζα και τα τεκτενόμενα στη Γάζα, αυτές οι διμερείς σχέσεις ε, έχουν διαλυθεί. Χρειάζεται να ανανεώσουμε το διάλογο. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Δεν μπορεί μόνο το Κοινοβούλιο ούτε η Κομισιόν να πούν την αλήθεια. Ο ρόλος των κρατών είναι πολύ αποφασιστικός. Αλλά ίσως μπορούμε να στραφούμε προς το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για να υπενθυμίσουν στα κράτη ότι είναι υπόλογα για τις αρχές που προωθούν και είναι υπόλογα για το κοινό μας μέλλον στην Μεσογειακή περιοχή. Γιατί αν είναι κάτι κρίσιμο σήμερα είναι ότι τελικά αυτό που κάνουμε είναι ότι προωθούμε τους πιο εξτρεμιστές ένθεν και ένθεν και ξέρετε ότι σε σχέση με ορισμένα δόγματα της άκρας δεξιάς του Ισραήλ Αυτά δεν είναι τα, τα μόνα ακροδεξιά λόγια που ακούμε και αλλού υπάρχουν ακροδεξιά δόγματα. Κύριε Έμερσον, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για τις, ε, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έχω να κάνω μια πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαλεία στη διάθεσή της απέναντι στο Ισραήλ. Και θα μπορούσε να πει ότι δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις ούτε νέα συμφωνία, νέα ανανεωμένη, αναβαθμισμένη συμφωνία, εάν δεν σταματήσει το Ισραήλ την επέκταση των επικισμών, αν δεν σεβαστεί το ανθρωπιστικό δίκαιο και αν δεν αφήσει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στα κατεχόμενα. Και να υποβάλουμε σοβαρές ειρηνευτικές προτάσεις για το θέμα της Ιερουσαλήμ και το χάρτη του Ισραήλ. Η κληρονομιά του Μπούς, που είναι αυτός ο κατάλογος των τρομοκρατικών οργανώσεων στα πλαίσια του πολέμου για την τρομοκρατία, σύμφωνα με όλους τους ανεξάρτητους αναλυτές, θεωρούν ότι είναι ένα απίστευτο αμάλγαμα η Χαμάς, ο Μπιν Λάντεν Η Βάσκοι, ο Ήρα, όλα ένας αχταρμάς. Και ήταν ε, ένα στρατηγικό α, λάθος και του Μπούς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησε. Έφυγε τώρα, ο Ομπάμα είναι πιο ανοιχτός. Και εμείς θα πρέπει να ξαναδούμε την αντίληψη που έχουμε για το ποιες είναι τρομοκρατικές οργανώσεις και ποιες όχι. Ευχαριστώ όλους τους ε, προσκεκλημένους για αυτή την ε, ενδελεχή συζήτηση που δεν οδήγησε σε προτάσεις, καινούργιες τουλάχιστον. Όλοι έχουμε τις αμφιβολίες μας, παρότι όπως ακούστηκε υπάρχει θέληση να προχωρήσουμε. Πολύ ωραία. Το δεύτερο τμήμα της ε, πρωινής μας συζήτησης αφορά ένα πακέτο από τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίας που συνδέονται και που αφορά τα, τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική περιοριστικών μέτρων ή κυρώσεων, τρεις εκθέσεις πρωτοβουλίας που συνδέονται, που εκπονήθηκαν από την Υποεπιτροπή σε αυτή τη διάρκεια, σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου Ζητήσαμε από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή να μας εξηγήσουν τις απαντήσεις, τις δράσεις δηλαδή που έχουν προωθήσει για να ληφθούν υπόψη αυτές οι συστάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λάβαμε το έγγραφο που μας έδωσε η Κομισιόν για το θέμα αυτό. Το Συμβούλιο μας είπε ότι δεν είναι σε θέση να μας στείλει γραπτή απάντηση για το θέμα αυτό. Η κυρία Κιόνκα όμως είναι εδώ και θα μας δώσει φαντάζομαι προφορικές απαντήσεις. Τώρα, πώς θα οργανωθούμε για αυτή τη συζήτηση. Ο καθένας από τους εισηγητές της έκθεσης, ο κύριος Ανιολέτο, ο κύριος Ομπιόλς και εγώ για την τελευταία έκθεση της κυρώσης, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας. Εν συνεχεία, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Αυνό και συνεχεία στην κυρία Κιόνκα. Και ξανά μετά στους βουλευτέ. Άξεχνα και την Προεδρία. Κυρία Ντουάζ, ε, καλημέρα σας και ζητώ συγγνώμη που σας παρέλειψα. Ο κύριος Ανιολέτο. Ξεκινάμε την πιο παλιά έκθεση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε εδώ, αλλά όχι μόνο που ήρθε, μόνο που ήρθε, αλλά και που έγραψε και ένα κείμενο και έδωσε λοιπόν συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα ήθελα να θέσω κάποια σημεία σε σχέση με τις παρατηρήσεις της Κομισιόν. Η Κομισιόν λέει ότι ετοιμάζει μια συνεισφορά που θα υποβάλει στο Συμβούλιο για τα σημαντικά σημεία του ψηφίσματος. Δηλαδή, το άρθρο του 96 που υπάρχει στη Συμφωνία της Κοτονού και το οποίο θα πρέπει να ενσωδιεθνεί συμφωνίες. Θα ήθελα να καταλάβω λίγο καλύτερα τι σημαίνει αυτό. Θα μπορούσατε να μας κάνετε ένα πρίβιο για αυτό το έγγραφο που ετοιμάζει η Κομισιόν ε, και που θα υποβάλει στο Συμβούλιο. Δεύτερον, η Κομισιόν λέει ότι θα διευρύνει το ρόλο των αρχηγών αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής, των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου, ούτω ώστε να κάνει σεβαστή ένα, μια ένα συγκεκριμένο αίτημα δηλαδή να έχουν μεγαλύτερο ρόλο οι αρχηγοί των αντιπροσωπιών ε, για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι σημαντικό νομίζω, γιατί η επιτόπια παρουσία επιτρέπει να παρατηρούμε ε, την κατάσταση όπως εξελίσσεται. Όχι να έχουμε μόνο μια, ένα στιγμιότυπο, ας πούμε, μια απεικόνηση, μια φωτογράφηση, αλλά να παρακολουθούμε την κατάσταση. Θα θυμάμαι, την ε, συζήτηση που είχαμε με τον αρχηγό της ε, Ευρωπαϊκής Αποστολής στην Κολομβία, που μου εξήγησε ποια είναι η κατάσταση. Θέλω να δω όμως ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος που θα αποδοθεί στους αρχηγούς των αντιπροσωπιών. Τρίτο σημείο. Μια μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση με τα στρατηγικά έγγραφα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι αυτό το σημείο είναι πολύ γενικό, λόγω δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Αυτό θέλω να το συνδέσω με κάτι άλλο, επί του οποίου δεν δόθηκε καμία πιστική απάντηση. Δηλαδή, στο ψήφισμα εμείς ζητούσαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε υποεπιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα έχουν και θεσμική παρουσία και θα βοηθήσουν ε, γενικά και τις οργανώσεις ε, και τις ευρωπαϊκές και τις οργανώσεις επιτόπου, ούτως ώστε να παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το Συμβούλιο Σύνθεσης θα ήθελα να προβλεφτεί η δημιουργία τέτοιων επιτροπών. Για αυτό το σημείο υπάρχει... δεν υπάρχει διάθεση. Επίσης, για το άρθρο 2 είχαμε ζητήσει τη δυνατότητα να αναδιατυπωθεί, γιατί μας φαινόταν τρομερά γενικόλογο. Επίσης δεν δόθηκε καμία απάντηση. Κάναμε αναφορά σε ορισμένε διεθνεί συμβάσεις. Παραδείγματο χάρη στη σχέση με την Τινησία. Υπάρχει ένα ολόκληρο θέμα με τους μετανάστες θα θέλαμε στις εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένες συμβάσει. Έτσι θα γινόμασταν πολύ πιο συγκεκριμένοι και όχι γενικοί και αόριστοι. Και επίσης δεν υπάρχει άνοιγμα της Επιτροπής. Μια τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξή. Υπάρχει και ένα ουσιαστικό πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, η διαχείριση είναι πάντα με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε για τη ρήτρα στις ε, συμφωνίες με την Κίνα. Το θέμα της εισαγωγής αυτής της ρήτρα ε, στη συμφωνία με την ε, Ινδία επίσης το έχουμε ξεχάσει. Ανάλογα με το πολιτικό και οικονομικό βάρος της ε, κάθε χώρας, ε, αποκτά διαφορετικό νόημα η ρήτρα. Και αν μια χώρα είναι, έχει το γεωπολιτικό βάρος του Ισραήλ, την ξεχνάμε τέλος τη ρήτρα. Επομένως, υπάρχουν σαφώς αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά ό,τι αφορά τη ρήτρα. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η γνώμη και του Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Γιατί, για να σας πω, γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις, ιδίω ό,τι αφορά τη συζήτηση για το άρθρο 96, η Κομισιόν πετάει το μπαλάκι στο Συμβούλιο και λέει ότι α, αρμόδιος είναι το Συμβούλιο. Σας παρακαλώ, ας μην πάμε από τον Αναστόν Καϊάφα. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη γνώμη έχει το Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ανιολέτο. Ο κύριος Ουμπιέλς, σε σχέση με την έκθεση για το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος και προσεκτικός γιατί πρόκειται για μια έκθεση την οποία δεν έχω συντάξει εδώ, εγώ, αλλά η συνάδελφος, πρώην συνάδελφος μάλλον, η Ελένα Βαλενθιάνο και εγώ απλώς παρακολούθησα την διαδικασία αυτή εκ των υστέρων συμμετέχοντας σε ορισμένες ε, συναντήσεις ενημέρωσης. Γι' αυτό θα περιοριστώ λοιπόν στο να κάνω καταρχήν ένα σχόλιο στην τελευταία παρέμβαση του Ανιολέτο και στη συνέχεια θα κάνω μια αξιολόγηση γενικής ε, φύσεως σε σχέση με αυτό που θεωρώ ότι υπήρξε η εξέλιξη της ε, ε, δράσης της Κομισιόν και του Συμβουλίου στην περίοδο μετά την έκθεση της κυρίας Ελένα Βαλενθιάνο. Χωρίς αυτό να σημαίνει μια αιτιακή σχέση μεταξύ έκθεσης και ε, κατοπινής εξέλιξης, γιατί πρόκειται για τέλος περίπλοκες εξελίξεις. Ο Ανιολέτο έχει δίκιο σε αυτό που λέει σε σχέση με την ε, χρήση διαμέτρων και σταθμών ε, και σε, σε πολλές περιπτώσεις. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την έκφραση που χρησιμοποιεί ένα ε, παλιός ε, φίλος μου συνδικαλιστή που αναφέρεται ε, συχνά στην ηλικιωμένη κυρία. Πώς είναι η ηλικιωμένη κυρία στην Γουατεμάλα ή πώς είναι η ηλικιωμένη κυρία στην Ιταλία. Και εγώ του, του ρώτησα, μα σε ποια ηλικιωμένη κυρία αναφέρεστε ε, και μου είπε στην, ε, στο συσχετισμό δυνάμεων. Αυτή είναι η γυραιά κυρία. Και η γυραιά αυτή κυρία ε, υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολο των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου έμεσα και της Κομισιόν και ίσως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν ε, η γυρά κυρία ήταν πιο δυναμική όσον αφορά την πράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, τα πράγματα θα ήταν ε, καλύτερα. Η γυρά αυτή κυρία λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει ο σχετισμός των δυνάμεων. Αυτό αφορά την ηθική και τις ε, ευθύνε ε, των πράξεων, όχι των αρχών. Αν η γυραιά κυρία δεν αλλάξει, όσο και ε, όποιες διακηρύξεις και να κάνουμε, ε, η πραγματικότητα δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν θέλω με αυτό να επικρίνω τον Ανενιολέτο. Θεωρώ ότι όσον αφορά την ουσία του θέματος, θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ θετικά την εξέλιξη των πραγμάτων σε αυτή την ε, περίοδο που ακολουθεί δηλαδή τον Οκτώβρη του 2007 όταν παρουσιάστηκε η έκθεση, όταν γκρίθηκε μάλλον η έκθεση Βαλανθιάνο. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη η οποία βασίζεται σε μια απόλυτη πεσιοδοξία, δηλαδή στη διαπίστωση του ποια είναι η κατάσταση ακριβώς της γεραιάς κυρίας, δηλαδή αυτού του σχετισμού δυνάμεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υπόλοιπο κόσμο, με τις μεγάλες δυνάμεις, με τις μικρές χώρες, με τα γεωπολιτικά προβλήματα, τα γεωστρατικά προβλήματα κλπ αλλά χωρίς αμφιβολία θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι σημειώθηκε μία εξέλιξη από ποσοτική άποψη θετική. Δηλαδή, ο αριθμός των διαλόγων ε, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι εμπιστευτικές ε, ε, συνεδρίες, οι, διοργανικές ενημερωτικές ε, συνεδριάσεις έχουν αυξηθεί. Όλοι οι εκπρόσωποι, η Κομισιόν, το Συμβούλιο κλπ. υπήρξαν διαθέσιμοι και επέδειξαν ένα πνεύμα συνεργασίας σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ε, χωρίς να θέλει κανείς, να μπορεί κανείς να θριαμβολογεί. Παρ' όλα αυτά έχουν σημειωθεί κάποιες πρόοδοι και σε θετική κατεύθυνση. Έχω την εντύπωση ότι πέρα από τις εκθέσεις και από τις συστάσεις των οποίων η εφαρμογή είναι αφισβητήσιμη, αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να επιδείξουμε μια θέληση διοργανικής εμπιστοσύνης, αν θέλετε. Ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Κομισιών, ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και αναφέρομαι στους κυρίους και κυρίες που στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο εργάζονται ακριβώς εδώ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί εδώ η γυραιά κυρία έχει μια πιο ευχάριστη όψη, δηλαδή ο συσχετισμός ε, δυνάμεων ε, είναι, μπορεί να αποβεί πιο θετικός και να πετύχουμε μια μεγαλύτερη συνένεση. Ευχαριστούμε κυρία, κύριο Μπιόλς. Είναι το θέμα κατά πόσο υπάρχει μια νομική ε, βάση για να υπάρξει μια τέτοιου είδους σχέση εμπιστοσύνης ή πίστης μεταξύ ημών. Η έκθεση για τις κυρώσεις ε, εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2008 Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν ε, ε, δεν έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα και οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από την Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, σε σχέση με τις στάσεις αυτές είναι περιορισμένες. Πρόκειται για μια έκθεση που αφορά τον εξορθολογισμό της πολιτικής επιβολής κυρώσεων, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνεπώς μεγαλύτερη αξιοπιστία. Πρώτη απαραίτητη δουλειά που αναφέρει και μια πρώτη σύσταση είναι να υπάρξει μια ενδελεχής ε, μελέτη επιπτώσεων, γιατί σήμερα δεν έχουμε καμία καθολική άποψη για τις επιπτώσεις των κυρώσεων που υιοθετούνται για καμιά τριανταριά χώρες. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα, μια μελέτη επιπτώσεων, σοβαρή μελέτη, για να δούμε πού βρισκόμαστε με τις κυρώσεις. Δεύτερον, να υπάρξει μια αυστηρή μέθοδος ε, με βάση κάποιες μελέτες με την αίσθηση ότι οι κυρώσεις είναι ένα εργαλείο πολιτικά ευαίσθητο και θα πρέπει να το χειριστούμε με γνώση, γνώση των συγκεκριμένων καταστάσεων των χωρών ε, που θα υποστούν τις κυρώσεις και θα πρέπει επίσης να έχουμε σαφή κριτήρια συγκεκριμένα ούτως ώστε να έχουμε μια θεώρηση από τη στιγμή που επιβάλλονται οι κυρώσει μέχρι τη στιγμή που θα έρθουν και με ποια κριτήρια θα έρθουν. Τρίτον, μια πολιτική κυρώσεων θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια μια συνολική πολιτική. Είναι ένα εργαλείο μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να συνοδευτεί και από μέτρα υποστήριξης της κοινωνία των πολιτών τη ε, εν λόγω χώρη, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μάχονται για να αλλάξουν κάποια πράγματα που υποτίθεται ότι αυτό θέλουμε και εμείς με την πολιτική κυρώσεων. Επίσης, διεύρυνση του πλαισίου ε, αιτίων που δικαιολογούν τις κυρώσεις, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την καταστροφή, τη ριζική καταστροφή του περιβάλλοντος. Το Συμβούλιο με έχει υποστηρίξει αυτό το σημείο. Η τελευταία μας πρόταση αφορά τη δημιουργία ε, ενός δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Γιατί πιστεύουμε ότι για να αποφασίσουμε το, τη φύση και το περιεχόμενο των κυρώσεων, ώστε να είναι αποτελεσματικές για κάθε περίπτωση, θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένα κριτήρια και να μπορούμε να προσμετράμε τακτικά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε να ενδυναμώσουμε την πραγματογνωμοσύνη που υπάρχει στην Κομισιόν, η οποία δεν έχει και πολλούς πόρους για αυτό το θέμα. Παρότι οι πόροι αυτοί είναι θαυμάσιοι, ε, δεν είναι αρκετοί για να κάνουν αυτή την τόσο περίπλοκη δουλειά. Ανθρώπινοι πόροι και, άλλα, και άλλοι. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει αυτό το δίκτυο των εξάρτων εμπειρογνωμόνων για να υποστηρίξουν αυτή την πολιτική των κυρώσεων. Αυτέ είναι οι βασικέ συστάσει τη ε, έκθεση για τι κυρώσει. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Αγνό, η οποία είναι η αγαπημένη μας ε, διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κυρία μου, σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα, γιατί έχουμε στείλει και αυτό το κείμενο, όπως, είπατε. Είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε από κοινού αυτές τις εκθέσεις, Γιατί μία από τις προκλήσεις που έχουμε σε αυτό το τομέα είναι η συνέπεια. Πώς θα είμαστε συνεπείς χρησιμοποιώντα όλα αυτά τα εργαλεία και πώς θα είμαστε συνεπεί παρεμβαίνοντα σε διάφορα επίπεδα. Για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, καλό είναι λοιπόν να εξετάσουμε από κοινού αυτέ τι εκθέσει. και σας ευχαριστώ που προβλέψατε κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε, ε, σε ό,τι αφορά το κείμενό μα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που μα είπαν οι συγγητές. Ο κ. Ανιολέτο θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα για τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε ό,τι αφορά την ε, συνεισφορά τη Κομισιόν. Δεν ξέρω αν είδατε ότι στην Κορεπέρ της 18ης Δεκεμβρίου του 2008 υπάρχει ένα ερώτημα που έγινε και προς την Γενική Γραμματεία και προς την Κομισιόν να γίνει ένα κοινό έγγραφο για να δούμε, να κάνουμε ένα απολογισμό αυτών των ρητρών. Σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όλοι συμφωνούν ότι είναι μια ρήτρα πρίμους ε, interpares, ε, βασίζεται στη συνθήκη, υπάρχει σε όλες τις συμφωνίες και θα παραμείνει και συνδέεται με μια ρήτρα αναστολής μια ρήτρα αναστολή η οποία επιτρέπει σε έκτακτες περιπτώσεις να λάβουμε μέτρα που μπορούν να φτάσουν, που είναι μέτρα έκτακτα καταρχήν, προσωρινού χαρακτήρα και θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το κοντονού ως παράδειγμα για να συστηματοποιήσουμε τη χρήση αυτών των ρητρών και να είμαστε σε καλύτερη θέση απέναντι στους εταίρους μας για να μην υπάρχουν τεράστιες διαφορές ως προς τον τρόπο που τους μεταχειριζόμαστε. Επομένως χρησιμοποιούμε το, τις ε, συμφωνίες μοντέλο. Δηλαδή, μια συστηματική έκτακτη διαβούλευση με όλες τις χώρες όταν χρειάζεται. Όλοι αυτοί, ε, όλοι στηλιτεύουν τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά εμείς την έχουμε στη βάση της πολιτικής μας, που θα πρέπει, θα πρέπει η πολιτική μας να έχει και συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, οι χώρες να ζητήσουν τις χώρες να επικυρώσουν τις διεθνείς συμβάσει καταρχά. θα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να προωθήσουμε προγράμματα που χρηματοδοτούνται εν μέρη από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθηθούν ε, κάποια στοιχεία πολιτικής. Εδώ και πέντε χρόνια βλέπω ότι υπάρχει ένας προτασιασμός ρητρών πέρα από την ρήτρα αυτή. Ε, αυτό το κείμενο λοιπόν που κάνει τον απολογισμό των ρητρών ετοιμάζεται από την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τους αρχηγούς των αποστολών και αντιπροσωπιών της Κομισιόν. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους. Ε, σημαντικός ο ρόλος και της Κομισιόν αλλά και των κρατών μελών. Η Κομισιόν έχει γραφεία ή μάλλον αντιπροσώπηση παντού, ενώ τα κράτη-μέλη όχι παντού. Σε ό,τι αφορά του αρχηγού των αποστολών, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη εντολή. Το ανέφερε και η κυρία Φλότ. Έχουν μια υποχρέωση στα πλαίσια του ρόλου του political reporting να κάνουν εκθέσει για τα ανθρώπινα, ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή έχουν επίση υποχρεώσει να έχουν τακτικέ επαφέ με την κοινωνία των πολιτών και μαζί με τους συναδέλφους των ε, πρεσβειών των κρατών μελών έχουν μια υποχρέωση μία φορά το χρόνο να κάνουν μια γενική έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πριν από κάθε διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάνουμε επίσης ένα απολογισμό. Επίσης, μαζί με την Τσεχική Προεδρία κάναμε κάτι που ήθελε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσπαθήσαμε να διαρθρώσουμε τον διάλογο που είναι πολιτικός και τα εργαλεία που είναι εργαλεία συνεργασίας της Κομισιόν και των κρατών μελών. Και ζητήσαμε από τους επιτόπιους αρχηγούς πριν από τις ε, επαφές που θα κάνω με τις τρίτες χώρες να μας δώσουν ένα κατάλογο προγραμμάτων και σχεδίων και να μας κάνουν και μια ποιοτική αξιολόγηση. Θα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των αρχηγών των αποστολών. Ε, έχουμε αποκεντρώσει την εφαρμογή της βοήθειας στο όσο μπορούμε περισσότερο. Βασιζόμαστε δηλαδή στο, στους αρχηγούς των αντιπροσωπιών με πολύ έντονο τρόπο. Συχνά ε, αυτοί κάνουν εκκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκκλήσεις που προσαρμόζονται στην κατάσταση που υπάρχει επιτόπου. Επίσης, ε, στα πλαίσια της συνένεσης για την ανάπτυξη θα πρέπει να δούμε ποιος κάνει τι για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Επίσης, μαζί με τους βασικούς διεθνείς δωρητές ε, και με τις υπηρεσίες του ΙΕ να, να δουν τι συμβαίνει. Ε, τελευταία, κάνουμε πολύ πρόοδο ό,τι αφορά κάποια συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις γυναίκες και τα παιδιά. Ε, ανταλλάξαμε επιστολές με τη UNICEF και με την UNIFAM, ούτω ώστε να υπάρχει συνεργασία με τις αντιπροσωπείες μας με σκοπό την αποτελεσματικότητα. Επίσης, μιλήσατε για κάτι που σας ενοχλεί σε ό,τι αφορά αυτό το έγγραφο στρατηγικής για τις χώρες ε, ότι δεν είμαστε πιο συγκεκριμένοι δηλαδή, αυτό μας κατηγορείται. Γιατί, Γιατί αυτή τη στιγμή ε, επανεξετάζουμε αυτά τα έγγραφα στρατηγικής αναχώρα. Εγώ θα ήθελα να δούμε τι προτεραιότητες έχουμε. Σε ό,τι αφορά ε, το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, έχουμε έξι διαλόγους Τρόικα, συν ε, του Ιράν που έχουμε σταματήσει το διάλογο, μαζί με το συνάδελφο από την Προεδρία και τον εκπρόσωπο του κ. Σολάνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, έχουμε έξι συμβουλευτικές τρόικες μαζί με τη Ρωσία. Δηλαδή, διαβούλευση τι σημαίνει. Ε, ποτέ ήταν οι χώρες που είναι πιο κοντά μας, πιο ανεπτυγμένες αν θέλει, πιο κοντά σε εμά. Από τις, τους 30 διαλόγους. Έχουμε 14 υποεπιτροπές ε, ε, συμφωνιών σύνδεσης, συμφωνίες που διαπραγματεύτηκε η Κομισιόν και έχουμε τρεις διαλόγους σε τοπικό επίπεδο που είναι εξελίξη. Βιετνάμ, Πακιστάν, το λέω γιατί αναφέρεται την Ινδία. Και επίσης ε, και με την Αρμενία, Γεωργία και Αζερβαϊτζάν ε, έχουμε διάλογο αυτό το εξάμεινο στα πλαίσια της Τσεχικής Προεδρίας. Έχουμε πολλά πράγματα να εξελίξει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, σε αυτά τα έγγραφα στρατηγικής αναχώρα θα θέλαμε να δούμε τις προτεραιότητες, τόσο ώστε να πούμε, αυτό το θέμα για αυτή τη χώρα είναι προτεραιότητα. Γιατί λέμε ότι το θέμα γυναίκες ή παιδιά μας ενδιαφέρουν ε, ή γιατί έχουμε ένα διάλογο. Θα προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε τα μεν τα δε. Ε, παρότι η εντολή για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορά όλους τους αρχηγούς ε, αποστολών, δεν θα το βάλουμε ως προτεραιότητα σε όλα αυτά τα έγγραφα στρατηγικής. Γι' αυτό δεν σας απαντάμε τώρα, γιατί το ξαναβλέπουμε μαζί με τους συναδέλφους αυτό το θέμα. Το θέμα είναι δηλαδή να έχουμε περισσότερη ε, αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα παραδοσιακά γεωγραφικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο κύριος Ομπιόλς μίλησε για την έκθεση ε, Βαλενθιάνου και μίλησε για δύο σημαντικά θέματα. Είπε ότι ε, ε, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και ναι και όχι. Είναι σαφές ότι στις εξωτερικές σχέσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή είναι μία από τις αξίες μας και επειδή είναι ένα πράγμα που μας χαρακτηρίζει, είναι κάτι που το βλέπω μακροπρόθεσμα. Αλλά έχουμε και άλλα συμφέροντα. Είναι προφανές δηλαδή ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Κίνα για την Γερμανία με τον ίδιο τρόπο. Είναι θέμα πολιτικό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε συστηματικοί με όλες τις χώρες. Φυσικά, ε, σε πολιτικό επίπεδο υπάρχουν διαιτησίες που προχωράνε, αλλά τίθενται και κάποια θέματα με βάση συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμές ε, για το τι θα θέσουμε στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν είναι για όλε τι χώρε το ίδιο. Θα πρέπει επίσης να δούμε τα πράγματα μέσα στην εξέλιξή του. Ε, εμείς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε μέσα σε 400 χρόνια και παρόλα αυτά έχουμε ακόμα πολλά εσωτερικά προβλήματα. Ε, συχνά παίζουμε πινκ-πονγκ με τους Ρώσους και με άλλους, ε, οι οποίοι μας λένε «Κοιτάξτε τι γίνεται στη δική σας ε, επικράτεια, μην μας κατηγορείτε εμάς». Ε, θα πρέπει να δούμε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα σε, σε μια εξελιχτική πορεία. Δεν μπορούμε να ε, λέμε ότι δεν πάει τίποτα καλά στην Κίνα. Η Κίνα έκανε θαυμάσια πράγματα μέσα σε 30 χρόνια. Έκανε τεράστια βήματα. Αυτό που θα ήταν καταστροφικό θα ήταν να μην υπάρχει καμία εξέλιξη και για μένα και για την Επίτροπο. Ε, από εκεί ξεκινάει ο διάλογος. μια χώρα η οποία αρχίζει τώρα να ανοίγεται δεν μπορεί να έχει το ίδιο επίπεδο με εμά. Αυτό είναι προφανέ. Το θέμα είναι πραγματικά δύσκολο. Ε, δεχόμαστε τι κριτικέ. Ε, Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε συστηματικοί και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ε, και, και εσείς κύριε Μπιόλης αναγνώρισατε ότι υπάρχουν θετικά θέματα. Ε, κάποιοι συνάδελφοι, όπω η κυρία Κιόνκα, που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, θα σα επιβεβαιώσουν ότι πραγματικά έχουν σημειωθεί πολλά βήματα προ τα εμπρός. Σε πολλού από αυτούς τους διαλόγους. Ε, οι διάλογοι αυτοί δεν είναι ένας σκοπό. Το γεγονό ότι υπάρχουν όλο και περισσότερε χώρε με τι οποίε κάνουμε αυτό το διάλογο και που αισθάνονται υποχρεωμένε να μα απαντήσουν, καλό σήμα είναι, καλό μήνυμα είναι. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα θέματα Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά τη θανατική ποινή και σε ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών και των παιδιών. Αυτά τα δύο θέματα. Δύσκολα βέβαια να κάνουμε μια σωστή αποτίμηση. Ένα από τα αιτήματα του Συμβουλίου για το διάλογο της Τρόικα είναι να κάνουμε καλύτερο, απολογισμό, καλύτερη αποτίμηση. Θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι προκλήσεις που αναφέρονται στην έκθεση του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α, κυρία Φλότ, ξέχασα να μιλήσω για τις κυρώσεις. Και οι κυρώσει είναι μία από τις ε, επικρίσεις που δεχόμαστε, ότι εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο στις σχέσεις μας. Υπάρχουν διαιτησίες, υπάρχουν εργαλεία της ΣΚΕΠΑ, σε ό,τι αφορά το δίκτυο των εμπειρογνωμόνων. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο σε επίπεδο κομισιών. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μελέτες για να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις και τι διαφορά έχουν οι κυρώσεις γενικές και οι πιο συγκεκριμένες που αφορούν μια χώρα. γιατί θα θέλαμε να είμαστε συστηματικοί, θεωρητικός πώς. Αλλά εξορισμού αυτό το πρόβλημα είναι πολύ ιδιάζων, εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τι προκλήσει, υπάρχουν πολλέ. Καταρχά, να υπάρχει μια συνοχή, μια θεσμική συνοχή. Όλοι μας κερδίσαμε από την ύπαρξη αυτών των διαλόγων. Και είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε αυτό το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς ως θεσμικό όργανο. Υπάρχει πρόοδος αυτό. Σε ό,τι αφορά την ε, συνοχή μεταξύ των εργαλείων μεταξύ τους, σε... προσπαθούμε να προχωρήσουμε στις σχέσεις μας ε, κομισιών και κράτους μέλους. Επίσης, ε, να είμαστε συνεπείς σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Θεωρούμε ότι οι διάλογοι αυτοί είναι αμοιβαίοι διάλογοι. Αν έχουμε αμοιβαίο διάλογο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και αυτοκριτική. Δεν μπορούμε να κάνουμε κήρυγμα στους άλλους μόνο. Θα πρέπει να είμαστε πιστικοί ούτω ώστε να πείθουμε τις χώρες ότι είναι για το συμφέρον τους να σημειώσουν θετικά βήματα, να κάνουν πρόοδο. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν περισσότερη προσπάθεια στους κοινωνικούς και οικονομικούς διαλόγους. Ε, επιμείναμε πάρα πολύ για τα πολιτικά θέματα. Αυτή είναι μια μεγάλη κατάκτηση του 20ου αιώνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή. Αλλά για να προσαρμοστούμε περισσότερο στη γλώσσα των τρίτων χωρών θα πρέπει να είμαστε σε θέση και εμείς να δούμε τι κάνουμε στο εσωτερικό μας για να τους δώσουμε και καλά παραδείγματα προς μίμηση ε, να τους πούμε «Α, φυλακές, τι μπορούμε να κάνουμε, και εμείς έχουμε προβλήμα, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι, κατά πολέμηση των βασανιστήριων, μπλα μπλα μπλα». Αυτή είναι μια πρόκληση για όλα τα θεσμικά όργανα. Να δούμε τι γίνεται στον τομέα της ε, δικαιοσύνης και της ασφάλειας. Μια άλλη πρόκληση είναι το διμερές και το πολυμερές επίπεδο. Ακόμη και αν δεν φαίνεται, εμεί προσπαθούμε πολύ. Προσπαθούμε με την Λατινική Αμερική που ανέφερε ο κ. Σομπιόλ, γιατί τη γνωρίζει ιδιαίτερα καλά, προσπαθούμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να έχουμε ένα διάλογο στην Νέα Υόρκη και ένα διάλογο στη Γενέβη. Για να δούμε, έχουμε κοινά σημεία. Ε, πώς μπορούμε να διαρθώσουμε τον, το διμερές επίπεδο με το πολυμερές επίπεδο. Θα μπορούμε να πούμε ότι σε διμερές επίπεδο ε, υποστηρίζουμε ε, το να αποσυπρογράψουν οι τρίτες χώρε κάποιες συμβάσει και ταυτόχρονα προσπαθούμε για την θανατική ποινή, ξέρω εγώ, να προσυπογράψουν στις δικές μας, στα δικά μα ψηφίσματα κτλ. Επίσης υπάρχει για την κατάσταση των γυναικών, Υπάρχει το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 1325. Να το προσυπογράψουν χρειάζεται μια προσπάθεια, γιατί οι νοοτροπίες είναι διαφορετικές και τα θεσμικά επίπεδα ε, είναι διαφορετικά. Έχουμε τη Γενέβη και τη Νέα Υόρκη, εκεί παίζουμε σε διακυβερνητικό επίπεδο. Μια άλλη πρόκληση που έχουμε είναι το να έχουμε προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με όλους. Θα πρέπει να δούμε τι είναι πιο αποτελεσματικό και πού. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το mainstreaming, δηλαδή να κάνουμε να δούμε τι θέματα προωθούμε. Έχουμε όλες τις κατευθυντήρες γραμμές που είναι θεματικές, καταπολέμηση του βασανιστηρίου, θανατική ποινή, γυναίκες, παιδιά, να την διασταυρώσουμε με την διμερή στρατηγική. Ε, κατά περίπτωση όλα αυτά, παρά δεν σα ικανοποιεί. Μια άλλη πρόκληση είναι η κατάσταση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και θα τελειώσω με αυτό. Οι μη ΚΑΟ συνδέονται σε αυτό το διάλογο σχεδόν συστηματικά. Ε, είτε ο διάλογος είναι υπό μορφή Τρόικα, είτε ο διάλογος ε, υπό την αιγύτα της Κομισιόν. Με αρκετή επιτυχία. Προσπαθούμε όλο και περισσότερο να κάνουμε και τοπικό διάλογο αλλά με ορισμένε χώρε, όπω το Τουρκμενιστάν, α πούμε, δεν τα καταφέρνουμε. Προσπαθούμε, αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Επίση, ξέρετε ότι έχουμε αυτό το εργαλείο, που είναι το αγαπημένο παιδί του Κοινοβουλίου, που είναι ένα ενιαίο εργαλείο, μοναδικό εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που μα επιτρέψει. Μας επιτρέπει να συνεργαστούμε κατευθείαν με την κοινωνία των πολιτών. Βλέπουμε ότι η κοινωνία των πολιτών ε, έχει προβλήματα. Οι νομοθεσίε είναι αρκετά περιοριστικέ, η ελευθερία δεν υπάρχει. Είναι, και εγώ προσωπικά δεν ξέρω τι θα συμβεί με την οικονομική κρίση. Ε, βρίσκω θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχέση με αυτό το θέμα και νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα, ακόμα και το Κοινοβούλιο, όταν έχουν κάποιες επαφές θα πρέπει να εξηγούν ότι η υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανισμών τοπικών μη κυβερνητικών ενώσεων και αυτή είναι μια πρόκληση γιατί υπάρχουν οι μεγάλες κυβερνητικές οργανώσεις που είναι μεγάλες, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζουμε και τις μικρές τοπικές οργανώσεις που έχουν πολλές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα στο Κονγκό. Νομίζω ότι αυτό, αυτή θα είναι μια από τις πολλαπλές προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, για την υποστήριξή σας και όπως σας είπα, είμαστε απολύτως ανοιχτοί για να συνεχίσουμε το διάλογο με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αρνό για, αυτό το, για αυτά τα σχόλια και για αυτή την ε, πολύ ξεκάθαρη ανάλυση, πολύ κέρια ανάλυση. Η κυρία Κενκά έχει το λόγο. Κιονκά. Είστε ειδική εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυρίου Σολάνα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω καλύτερο είναι να μιλήσει η Προεδρία. si vous voulez. <laughs> Madame Doula. Kyria Doula. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την συνάδελφο από την Επιτροπή που μας έδωσε μια εξαίρετη επισκόπηση των ε, τριών ζητημάτων που αναφέρει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πράγματι θεωρούμε αυτές τις εκθέσεις πολύ σημαντικές και Κομισιόν με το Συμβούλιο θα δώσουν μια συνέχεια σε αυτές τις συστάσεις. Θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα βασικά σημεία στις δύο μάλλον αυτές εκθέσεις γιατί η Κομισιόν ήδη έκανε μια εξαντλητική παρουσίαση των συστάσεων που είναι μέρος ε, της έκθεσης για τις ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι η βασική ευθύνη της Κομισιόν ε, ε, του οργάνου εκείνου που εφαρμόζει και διαπραγματεύεται τις συμφωνίες αυτές. Να πω πρώτα απ' όλα πως το Συμβούλιο θα αρχίσει να δουλεύει σε αυτά τα πράγματα κατά την έκτη θητεία όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο πως πρέπει να αυξηθεί η συνοχή και διαφάνεια της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ένωσης και σε αυτό σκοπεύει και η τωρινή Προεδρία. Επίσης ε, Επίσης το αυξημένη έμφαση που πρέπει να δοθεί στην ε, δημοκρατία. αυτός είναι ο ένας στόχος που θα είναι στο κέντρο της ε, πολιτικής μας ε, και της ομάδας εργασίας. Όσον αφορά την έκθεσή σας για τις κυρώσεις, έχω να πω κάποια πράγματα. Οι βασικές αρχές για τις κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα βεβαίω αναφέρουν την ανάγκη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και βεβαίω πρέπει να η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα έχουμε ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως η διάσταση αυτή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε πως οι κυρώσει δεν εφαρμόζονται μόνο για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και για άλλου λόγους και στόχους όπως η ειρήνευση, η διεθνής ασφάλεια κέρια συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης, καθώς και η διεθνή συνεργασία. Οπωσδήποτε, η ομάδα εργασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασχολείται βέβαια με την τύχη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως ομάδα εργασίας θα συνεχίσουμε την πρακτική της Γαλλικής Προεδρίας να προετοιμάζουμε δηλαδή και να προσφέρουμε στις άλλες ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και στο Συμβούλιο γενικώ αξιολογήσεις ανά χώρα. Αυτό έγινε επί Γαλλικής Προεδρίας για το Ουσμπεκιστάν και θα αξιολογήσουμε τις πτυχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων των περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη Βυρμανία και τη Λευκορωσία στην επόμενη συνεδρίασή μας την ερχόμενη εβδομάδα. Επίσης, ε, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην κάθε χώρα και την άποψη άλλων φορέων αντί για την αξιολόγηση μόνο των Υπουργείων Εξωτερικών. Επίσης αναφέρθηκε ο ρόλος κοινωνίας των πολιτών επιτόπου στις χώρες αυτές. που τονίζουμε εμεί ω Προεδρία, αλλά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε οπωσδήποτε. Και αυτό είναι κάτι που υπήρχε σε όλους τους διαλόγους του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πτυχή δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών και συνεργασία. τονίζοντας πως οι κυρώσεις δεν έχουν πάντα μια λογική ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλό είναι με εδώ να τονίσουμε τον ρόλο της ομάδας εργασίας μας στο πλαίσιο αυτής της πολύπλοκης εικόνας που εμείς ως εμπειρογνώμονες σε αυτά τα θέματα προσπαθούμε να προωθήσουμε. Αλλά αυτό είναι ε, το πλαίσιο των πολύπλοκων σχέσεων με την κάθε χώρα. Όσον αφορά τις κυρώσεις, καλό είναι να πούμε πως ε, το Συμβούλιο εκτιμά την στήριξη του Κοινοβουλίου για την χρήση στοχευμένων κυρώσεων. Γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου και την ανθρωπιστική κατάσταση και τις συνέπειες στους πληθυσμούς και στις γειτονικές χώρες. Uh, uh, να καλωσορίσω επίσης ε, το γεγονός πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να φέρει αυτό το ζήτημα στις συζητήσεις με άλλες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε τη δυνατότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εξηγήσουμε στους εταίρους μας στον κόσμο το σκεπτικό της ε, πολιτικής μας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Επίσης χρήσιμο είναι να πούμε κάποια λόγια για τους διαλόγους γιατί κάνει διαλόγους η Προεδρία Οπωσδήποτε αυτούς τους οποίους κάνει η ομάδα εργασίας μας υπό τη μορφή και το σχήμα της Τρόικας και τους δομημένους μακροπρόθεσμους διαλόγους που κάνει εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία και την Κίνα π.χ. αλλά και διάλογο με χώρες π.χ. της Κεντρικής Ασίας ε, διάλογο που θα ξεκινήσει με τις χώρες του Νοτιού Καυκάσου. Χρήσιμο είναι νομίζω να πούμε πως μερικές φορές ο διάλογος όπως με την Κίνα ή την Ρωσία προσελκύει την προσοχή της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και λιγότερο ελκυστικοί διάλογοι ορισμένες φορές σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο και κλείνει το μικρόφωνο της Excuse me. Uh, yes, because some, some... Γιατί κάποιοι συνομιλητές μας θέλουν πιο πολύ να, έχουν, να έχει αποτέλεσμα αυτός ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση η ομάδα μας ε, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην περιοδική αξιολόγηση της χρησιμότητας των, του διαλόγου αυτού. Δεν αξιολογείται κάθε συζήτηση με τον ίδιο τρόπο, αλλά πάντα τονίζουμε στην σωστή συζήτηση το πώς θα ορίζεται η μερίσια διάταξη, να υπάρχει μια συνέχεια, να αντικατοπτρίζεται η κατάσταση στην κάθε χώρα, να συζητάμε κάποια σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε συνέχεια που δίνεται στο διάλογο. Προετοιμάζουμε επίσης ε, τον ε, κατάλογο θεμάτων που πρέπει να παρακολουθήσουμε και παρακολουθούμε μεταξύ των γύρων συνομιλιών ε, μέσω των αποστολών μας ε, στις διάφορες χώρες αυτά τα θέματα. Αυτή νομίζω είναι μια σημαντική πτυχή του πώς θα γίνει ο διάλογος πιο χρήσιμος και πιο αποτελεσματικός τελικά. Η Βερονή Καρνό τόνισε και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κρίσιμος προσπαθούμε να έχουμε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών από την κάθε χώρα συνεχώς ε, αυτό δεν είναι πάντα αποδεκτό από την άλλη πλευρά αλλά είναι κάτι το οποίο επιζητούμε και το θεωρούμε κεντρικό θέμα γιατί ο διάλογος πρέπει να γίνεται σε δύο επίπεδα και με τις αρχές και με την κοινωνία των πολιτών και με αξία της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της άλλης χώρας. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την τύχη να έχουμε εδώ την μελλοντική πρόεδρο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κυρία Μακόρτ, και θα σας δώσω το λόγο γιατί εσείς πραγματικά θα εξασφαλίσετε την συνέχεια, τουλάχιστον για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάποιων πρακτικών που έχουμε ξεκινήσει σε αυτή τη θητεία όσον αφορά τις διοργανικές σχέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων που μας δώσετε τη δυνατότητα. Ως ε, επόμενη Προεδρία, να πω πως ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας ε, κατά διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Και είπατε πως υπάρχει πράγματι η προοπτική της συνέχειας. Επί της ουσίας, η Προεδρία νομίζω εκπροσώπησε το Συμβούλιο Ε, αναμένω λοιπόν να συνεχίσουμε το διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κιονκά, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένε σύντομε ε, προσθήκες στα όσα είπε ε, Πρόεδρος του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Οι ρήτρε για τον ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομίζω ότι τονίστηκαν τα σημαντικά στοιχεία ε, υπάρχουν κεντρικές ε, ρήτρες, άλλες λιγότερο κεντρικές. Η συζήτηση η οποία γίνεται στο Κορεπέρ συνεχίζει και όπως είπε συνάδελφος από την Επιτροπή ε, συνεχίζεται αυτή η συζήτηση, είναι μια δεύτερη συζήτηση. Όσον αφορά την έκθεση Βαλενσιάνου, καταρχήν Ο κύριο Σομπιόλ έκανε μια θετική αξιολόγηση και συμφωνώ μαζί του. Νομίζω ότι ήρθαν πολλά θετικά στοιχεία από αυτή την έκθεση και από τις συζητήσεις ε, σχετικά με τις συστάσεις αυτής της έκθεσης. Ένα από αυτά είναι μια σειρά από εμπιστευτικά briefing τα οποία έγιναν με την Επιτροπή, τη Γραμματεία του Συμβουλίου και τους ε, ορισμένους ε, ευρωβουλευτές από αυτή την επιτροπή, που επιλέξαν από αυτή την επιτροπή. Και θα ήθελα να πω ότι εύχομαι στο μέλλον να υπάρξουν ίσως περισσότεροι βουλευτές που να δηλώνουν ενδιαφέρον για, αυτές τις εμπιστευτικές, ε, για αυτά τα εμπιστευτικά briefing, καθώς και για τις δημόσιες ακροάσεις που οργανώνουμε, όπως για παράδειγμα όταν μας καλέσατε να μιλήσουμε πριν ή μετά κάποιους διαλόγους σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτών των διαλόγων. Συνήθως υπάρχουν τρεις ή τέσσερις ε, βουλευτές και κανείς σχηματίζει την εντύπωση ότι είναι μόνο λιγοστοί αυτοί που ενδιαφέρονται για αυτούς τους ε, διαλόγους και θα είναι ωραίο να υπάρξουν περισσότεροι. Υπάρχει λοιπόν μια βελτίωση από αυτή την πλευρά των ε, πραγμάτων. Τώρα, ο κύριος Ομπιόλς επίσης αναφέρθηκε σε διάφορα τμήματα της έκθεσης και τις ανάγκες να υπάρχει μια διοργανική εμπιστοσύνη, να υπάρξει μια γέφυρα μεταξύ ορισμένων ατόμων. Δεν θα μπω στη συνέχεια συζήτηση για τη ρίση του Μοντεσκιό. Η κυρία Πρόεδρος την έχει ακούσει ήδη αρκετές φορές, αλλά θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων, όπως είπα, όπως είπα και όταν εγκρίθηκε αυτή η έκθεση για την αναφορά της ανάγκης να υπάρχει περισσότερο προσωπικό στη γραμματεία του Συμβουλίου σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πραγματικά θα ήταν καλό να υπάρχουν πιο συχνά τέτοιε αναφορέ, ούτω ώστε να υπάρξει μια αύξηση του δυναμικού, του προσωπικού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναφέρατε και πάλι. Τώρα, όσον αφορά τους διαλόγους, η συνάδελφος από την Επιτροπή μου υπενθύμησε ότι έχει νόημα να υπάρξει μεγαλύτερη επαγρύπνηση σε σχέση με το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει ένας διάλογος, υπάρχουν κατευθυντήριες ε, γραμμές για το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιπρόσθετα υπάρχουν και διάφορες άλλες κατευθυντήριες ε, γραμμές ε, για άλλα θέματα τα οποία βρίσκονται στις ημερήσεις διατάξεις διαφόρων διαβουλεύσεων με τις τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ και αυτό είναι το τρίτο σημείο εδώ, ότι τη διάρκεια των δύο τελευταίων προεδριών προσπαθήσαμε να αναθεωρήσουμε και να ανακαινήσουμε όλες ε, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επαναεξετάσουμε τη νέα κατευθυντήρια γραμμή για το ανθρωπιστικό δίκαιο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε τη μορφή ενός εγχειριδίου. Ε, ούτως ώστε να μπορεί να προσφυστεί ήδη το Μάρτιο, σε μια διοργάνωση Προεδρία το Μάρτιο. Έχουμε ανανεώσει λοιπόν όλες αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, έχουν όλες επαναπροσαρμοστεί τους τελευταίους μήνες από το Συμβούλιο. Τώρα όσον αφορά τις κυρώσεις, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ κυρία Φλότρ ότι η έγκριση αυτής της έκθεσης ε, έγινε πρόσφατα, συνεπώς είναι δύσκολο να, να αξιολογήσουμε την ε, δραστηριότητες ε, σε αυτούς τους διάμεσους μήνες. Το μόνο που θα μπορούσα να κάνω ή, να πω είναι ότι θα ήμουν κάπως απρόθυμη στο να υποστηρίξω μια άποψη σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένας υπερβολικός αυτοματισμός στο σύστημα γιατί μειώνεται ο ρόλος των πολιτικών και των πολιτικών αποφάσεων και αυτό είναι ένα θέμα, είναι σειρά της, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από το Συμβούλιο. Νομίζω ότι οι πολιτικοί προβληματισμοί θα πρέπει να διαματίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ. Και νομίζω θα περιοριστώ εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά λέει περίπου η εκθέσή μου. Θα έπρεπε να το διαβάσετε, γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Υπάρχει κάποιος βουλευτής που θέλει να πάρει το λόγο. Ο κ. Σανιολέτο, ο κ. Σομπιόλς. Ε, να ανταπαντήσει αυτά που απάντησε το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Ο Σανιολέτο. Eh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν γιατί ε, έκανε μια προσπάθεια καημένη για να μπει στην ουσία του θέματος. Ίσως πιο χρήσιμο θα ήταν να δούμε καταρχάς πιο συγκεκριμένα το, το κείμενο της Κομισιόν για να δούμε και πώς εφαρμόστηκε αυτή η ρήτρα. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Συμβουλίου, τι να σας πω κυρία μου, δεν ξέρω τι να σας πω. Ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ότι πρέπει να συνεργαστούμε, συνεργαστούμε ότι πρέπει να υπάρχει συνέχιση των προσπαθειών των προδριών δεν χρειάζεται να έρθει κανεί στο κοινοβούλιο για να τα μάθει. Τα παιδάκια που έρχονται από τα σχολεία εδώ τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Έτσι όπω είναι η θεσμική αρχιτεκτονική τη Ευρώπη για αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν μπορεί να κινηθεί μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, μέχρι να υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έχει εκτελεστική εξουσία. Από αυτή την άποψη. Δεν μου δώσετε καμία απάντηση, κυρία μου. Ούτε καν για το πρώτο σημείο. Τη εφαρμογή του άρθρου 96. Το θέμα τη ε, δυνατότητα διμερού άρση ε, των συμφωνιών. Τι γνώμη έχει το Συμβούλιο. Δεν έχει... Για την επίσημη εμπλοκή των, επιτρο... των υποεπιτροπών. Δεν μου δώσετε καμία απάντηση. Η Κομισιόν ανέφερε διάφορα προβλήματα επί των οποίων μπορούμε να συζητήσουμε. Τι να σας πω λοιπόν. Περιορίζομαι να πω ότι αν εδώ έχουν φτάσει τα πράγματα, ε, το επιτρέψω μια τελευταία παρατήρηση. Και στις ε, ετήσιες εκθέσεις που γίνονται από το Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προσέγγιση μας δεν είναι το να συζητήσουμε μόνο κατά περίπτωση. Να πούμε ότι για αυτού τους έξι μήνες η Προεδρία διάλεξε τρεις χώρες από τις 40 ε, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Εντάξει, αυτή είναι μια επιλογή με πολιτικά κριτήρια. Το δικό μας πρόβλημα δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Μέσα στην ε, γενική οικονομία, των στην γενική αρχιτεκτονική που υπάρχει, κάναμε συνολικά βήματα προς τα εμπρός για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε να έχουμε ε, ρήτρε που εφαρμόζονται πάντα, δεν εφαρμόζονται αυτόματα και να ξέρουμε ότι υπάρχει πρόοδος. Επί των συγκεκριμένων σημείων το Συμβούλιο δεν είπε τίποτα. Δεν μου είπε τίποτα για το άρθρο 96. Δεν μου πει τίποτα η Προεδρία. Είμαι εντελώς ανικανοποιήτο από την απάντηση του Συμβουλίου. Αν συμφωνεί και η Πρόεδρος, θα ήθελα να του ζητήσουμε ε, ένα γραπτό σημείο. Γιατί όταν μας στέλνουν ένα κείμενο, να μας στείλουν ένα γραπτό κείμενο. Γιατί όταν μα θέλουν κείμενο δεν μπορούν να είναι τόσο γενικοί και αόριστοι. Να έχουμε κάτι επί του οποίου να συζητήσουμε τέλο πάντων. Ναι, μα αυτό ακριβώ κάναμε, είπαμε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να μα απαντήσουν ε, γραπτά. Δεν έχουμε όμως τίποτα από το Συμβούλιο, έχουμε από την Κομισιόν. Ε, περιμένουμε λοιπόν κάποια στοιχεία απάντησης από το Συμβούλιο, τα οποία να είναι πιο ακριβή σε σχέση με διάφορα στοιχεία συστάσεων που περιλαμβάνονται στις τρεις μας εκθέσεις. Κύριε Μπιόλ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι. Ωραία λοιπόν. Τότε σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα κλείσουμε εδώ τη συνεδρίασή μας. Ε, μια και δεν θέλει, δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω και δεν θέλει και κανείς να πάρει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, εν πάση περιπτώσει, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διάφορους εκπροσώπους του Συμβουλίου και την κυρία Κιονκά για την παρουσία τους εδώ.